Good afternoon. Γεια σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Please take your seats. And please get ready. Λοιπόν, βλέπω κάτι συντονιστές ακόμα να εργάζονται επί σκηνής, ζωντανά, για να ολοκληρώσουν τον κατάλογο ψηφοφορίας για ποια έκθεση όμως. Λοιπόν, περιμένουμε άλλο ένα λεπτό να ολοκληρώσουν οι συντονιστές το συντονισμό τους. Εσείς έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες και περίπλοκες αρκετά. Λοιπόν, προπάσεις άλλης εργασίας, δοκιμάστε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Παρακαλώ. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Can you can you can you ask your assistant to get for another one? To I mean to fetch another one, to fetch a new one. It'll take some minutes, but we in the meantime we Λοιπόν, στο μεταξύ θα σας μετράμε κυρία Παπαδοπούλου όταν σηκώνετε το χέρι σας. Ε, αρχίζουμε λοιπόν. Καθίσατε όλοι είστε έτοιμοι, πάμε. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι Έχουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Μια σειρά ψηφοφοριών και αμέσω μετά θα ψηφίσουμε μια έκθεση αρκετά περίπλοκη της κυρίας Φλασίκο Βαμπένοβα. η οποία είναι μακροσκελής έκθεση και πολλή δουλειά μας περιμένει. get started with the first Αρχίζουμε λοιπόν πρώτη ψηφοφορία. Ε, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα Ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα. Εισηγητής είναι ο κύριος Τίμωθη Κίρκοπ. Θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Σιγητά, αν όχι να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Τώρα δηλαδή. Πέρασε. Έληξε. 31 υπέρ, 18 αποχές και μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση του κυρίου Κίρκοπ. Ευχαριστώ πολύ. I understand the commission. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι κατάλαβα, βάσει του αποτελέσματος θα ήθελε να λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λιγότερο από ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της ε, και ε, τη θλίψη της για την ε, έκβαση αυτής της έκθεσης. Η μελέτη που προτείνουμε είναι η απάντηση από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και των εμπειρογνωμόνων για ένα πρόβλημα ε, που φιλοδοξούσε να καταγράψει τον ευάλωτο πληθυσμό που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ακολουθήσαμε τις ε, ε, συστάσεις του ΟΗΕ, έχουμε πυρογνώμονες, άρχισε το πακέτο από τη Χάγη και συνεχίστηκε στη Στοχόλμη και το Συμβούλιο ήδη είχε βρει ε, ειδική πλειοψηφία για να υπερψηφίσει αυτή την πρόταση. Και για να τελειώσω, ε, λυπάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν μπορεί να μπει σε αντίστοιχη συζήτηση τώρα με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Okay, Μάλιστα. Καλώς ε, το πήραμε το μήνυμα ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σημειώνουμε. Το μήνυμα ελήφθη. Έκθεση Δάνοκα. Έχουμε και ψηφοφορία για την έκθεση Στάντλερ, αλλά δεν πρόκειται πλέον ε, να ψηφιστεί, έχει καταπέσει ε, λόγω της προηγούμενης ψηφοφορίας. Ερχόμαστε στην έκθεση Στάνοκα, πολιτές πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης για την περίοδο 2013-2017. Και εδώ πάλι ε, ακούμε... Α, ψήφι υπέρ, η συγγήτρια τι λέει. Κυρία Στάνοκα, ορίστε, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή μας ε, Πολιτικών Ελευθεριών μια στρατηγική για την έκθεση αυτή. Έχουμε ήδη συζητήσει ε, σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και με τους σκιώδεις ηγητές και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου θα πρέπει να δώσουμε ε, την συνένεσή μας έστω και απρόθυμα διότι θα πρέπει να λειτουργήσει ε, ο Οργανισμός Εμελιωδών Δικαιωμάτων μετά την 1η Πρώτου 2013. Ακόμα και αν είναι φιλόδοξη η εντολή της, Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε όμως στο Συμβούλιο ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μπορεί το Βρετανικό Κοινοβούλιο ε, να καθυστερήσει μήνες να εγκρίνει την εντολή. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το εξής ως τακτική. Να εγκρίνουμε πρώτα την έκθεση αυτή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Μετά, αν έχουμε καλά νέα από το Συμβούλιο, να ξαναφέρουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια πριν την ψηφοφορία για να επανέλθει το Συμβούλιο και να κάνει τη δήλωσή του. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει πρόοδος, να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και να ζητήσουμε δήλωση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια με συζήτηση και ενδεχομένως ψήφισμα. Αυτή είναι η πρότασή μου στην Επιτροπή και όλοι οι σκιώδεις επαναλαμβάνω συνεφώνησαν. Okay. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Το σημειώνουμε και αυτό. Τι ζητάτε λοιπόν. Υπάρχει τελική ψήφος για το σχέδιο ε, σύστασης, αλλά θα κάνουμε δύο, όχι δύο ψηφοφορίες, μία ηλεκτρονική ψηφοφορία αρκεί. Ψηφίζουμε λοιπόν αμέσως για το σχέδιο της σύστασης ηλεκτρονικά, αρχίζει ψηφοφορία. Και τελειώνει. Α, ένα σοσιαλιστή παραπάνω. Η κυρία ε, Παπαδοπούλου έχει την κάρτα τη. Θα τη φέρει βοηθό μου. Υπερψηφίζω όμω. Ωραία. 43 υπέρ, καμία αποχή και 11 κατά. Ε, σημαίνει ότι εγκρίνεται το σχέδιο της σύστασης. Συγχαρητήρια κυρία Σδάνοκα. Και τώρα ερχόμαστε στην ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συγκήτριά μας είναι η κυρία Μόνικα Φλασικόβα Μπενοβά. Εδώ ανακοινώνω ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας είναι 50 σελίδων. Κόλαση, σκέτη δηλαδή. Οπότε ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για τα αναπόφευκτα λάθη που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν. Κυρία Φλασικόβα, θέλετε να πείτε τίποτα. Όχι, αρχίζουμε. Then, the situation, the situation is good enough. Λοιπόν, έχει ε, κατάσταση αρκετά καλά. Αρχίζουμε. Η τροπολογία 58, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε να το ελέγξουμε. Τι ελέγχουμε. Την 62. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 29 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. Τώρα, ναι, έχετε την κάρτα σας. Όχι ακόμα. Συμβαστική 1α υπέρ, κατά. Abstentions adopted. 63 favor. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές ε, εγκρίνεται. 64 ήταν αυτή. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 και 72 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 68 κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Το τρίτο υπέρ Α, ζητώ συγγνώμη, είχε εγκριθεί, λέει ο πρόεδρος. Άρα καταπίπτει. Όχι, τώρα πάμε στο τέταρτο, γιατί το τρίτο καταπίπτει. Κατρία παχτή στα γαλλικά. Είπε. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, παρακαλώ επαλήθευση. Για το τέταρτο τμήμα της 68 αρχίζει τώρα. Πέρας. 29-25. Εγκρίνεται. Σημεία 30. 25. Συμβαστική τροπολογία 2. Επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 Επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 73 Επέ. Κατά. Αποχές απορρίψετε Η 76 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Ναι. Νομίζω ήταν ίδια πλειοψηφία πριν από λίγο, αλλά ας το ελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 76. Πέρας. 29-26. Συν την κυρία Παπαδοπούλου 30-26. Η 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα που πάμε στην 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Α, τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Α, ίδια πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα, το πρώτο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, 29 προς 24 και ξανά το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. «91. Έλεγχος ηλεκτρονικός παρακαλώ της 91. Άρχεται η ψηφοφορία». Πέρας ψηφοφορίας. 28 έναντι 26 δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 και 96 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβιβαστική 4 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή τον 6 πρώτη πρόταση. Μόνο την πρώτη πρόταση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερη πρόταση. Όχι. Α, καταπίπτει. Προχωρούμε στην 110. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 111 και 112 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 αποσύρεται. 115, 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δεκαεννέα, εκατόν είκοσι, εκατόν είκοσι ένα είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 122. Πρώτο τμήμα. Είναι ε, κατά τμήμα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 127 έχει αποσύρεται 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ. Κατά. Α, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε? 100, της 141. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Την 141. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 145, 46, 47. Α, 145 και 146 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Ε, είναι, δεν είναι ε, σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. 145-146. Πέρασε τη ψηφοφορία. 23 ψήφοι έναντι 33 απορρίπτονται. Απορρίπτονται. Είναι λοιπόν σίγουρο το αποτέλεσμα με το ηλεκτρονικό τσεκάρισμα, όχι με την ε, ανάταση των χεριών. Αλλά παρακαλώ όταν σηκώνετε το χέρι σας ε, να βλέπουμε καθαρά. 147 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Α, το τρίτο τμήμα καταπίπτει, εφόσον εγκρίθηκε το δεύτερο. 155, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 156, 157, ε, ταυτόσημες, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται, 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 100 Οι επόμενες δύο έχουν καταπίπτουν. Προχωρούμε ε, συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168. Υπέρ. Κατά. Μάλλον καταπίπτουν, καταπίπτουν. Ρωτάει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, καταπίπτουν. Οπότε προχωράμε... Α, πρέπει να ψηφίσουμε όμως. Πρέπει. Την 168 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, 177. Υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 178. Ε, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 179. 178. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ελ, ε, πέρας της 22 έναντι 33. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184-85 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 δεύτερο τμήμα δεύτερο τμήμα της 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 195. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 22 έναντι 34 απορρίπτεται, απορρίπτεται. Γι' αυτό παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201-202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 217 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το 31 24 εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 223 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 226-224 είναι ίδιες, υπέρ. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική πρόταση 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ. Και 230 που είναι ίδιες, ταυτόσιμες. Α, δεν είναι, δεν είναι, όχι. 228. 228 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 230 και 231 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται, 232 υπέρ, κατά, ας το επαληθεύσουμε για την 232, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 30 με 27. Υιοθετείτε. 233 υπέρ. Κατά. Το επαληθεύουμε ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 28 με 27. Υιοθετείτε. Οι 234 και 35 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 236 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, 237, η 238 είναι ταυτόσιμες, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική πρόταση 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε για την 245. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23 με 34 απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχέσα. Υιοθετείται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249, ξεχωριστή ψηφοφορία, ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο κομμάτι, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε για το δεύτερο κομμάτι. 249 επαληθεύουμε την ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 33, 32 ε, συγγνώμη με 24. Εγκρίνεται. Πάμε στο διεθνή 250. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία για το 252. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Το πρώτο κομμάτι... Να το διαβάσω? Όχι. Όχι, από εκεί επαναλαμβάνει rates until services. Είναι το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι είναι in some member states macro family planning. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι από το rates, Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο κομμάτι, υπέρ, κατά. Λοιπόν, ας το τσεκάρουμε, ας το επαληθεύσουμε, συγγνώμη. Για το δεύτερο κομμάτι. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 με 23. Εγκρίνεται. Πάμε στο 250, στην 253. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 258 ξεχωριστή ψηφοφορία, το πρώτο κομμάτι, υπέρ, Πρώτο κομμάτι είπαμε. Α, έχει εκπέσει. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπέρ. Α, και αυτό καταπίπτει. 259 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 260 και 61 ταυτόσημες, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 263-64 ταυτόσημες, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 265 και 66 ε, και 67 ε, ταυτόσημες υπέρ, πρέπει να... Λοιπόν, ψηφίζουμε την 265 όμως πρώτα. Πρώτα την 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, 266 και 267 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 268. Υπέρ. Κατά. 269 με, με προφορική τροπολογία υπέρ. Έχει απορριφθεί, έχει απορριφθεί ή όχι. Όχι, μάλλον έχει καταπέσει ή όχι, συγγνώμη. Να ψηφίσουμε ή όχι. Επιμένει κανείς να ψηφίσουμε. Όχι. Αποσύρεται. 270. Ξεχωριστή ψηφοφορία. 270 το πρώτο κομμάτι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο κομμάτι. Υπέρ. Ε, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 271 ξεχωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ε, παληθεύουμε το δεύτερο κομμάτι. Άρχεται η ψηφοφορία. Now 26 Λοιπόν, 32-26 εγκρίνεται. 271. Έχει καταπέσει. Όχι. Εντάξει, δεν το ψηφίζουμε. 272 και 273 και 274 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 275. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουν το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Against. Abstentions. Adopted. Εγκρίνεται. 276. 276. Α, έχει καταπέσει. 277 και 278 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, 279 το δεύτερο κομμάτι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 280. Υπέρ, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο τμήμα. 280 το πρώτο τμήμα. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 282, 282 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 285 και 286 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 291-292 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 293-94 και 96 και 97 όχι όχι. 293 και 294 μαζί, μαζί, τσουζάμεν οι 96, 293 και 94, Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, οι 296 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 297. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 295, 300 και 305. Και 305, αν δεν κάνω λάθος, είναι μαζί και οι τρεις, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 306 και 308, πάλι μαζί, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 310 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 311 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 313 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 314 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 316 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 317 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 318 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 319 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 320 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική πρόταση 21 υπέρ, κατά αποχές Υιοθετείται 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 όχι, όχι και αυτή, καταπίπτει επομένως πάμε στη βασική πρόταση τη συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 332 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 333 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 342 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 345 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 347 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 349 όχι 348 348 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 351 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 352 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 354 υπέρ κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 που πάμε τώρα μια στιγμή 372 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 373 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 378 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 381 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 392 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 393 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη έχει αποσυρθεί 395 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 400 και 401 ευτυχώς απεσύρθησαν και πάμε στη 402 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 403 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 404 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 409 Υπέρ. Κατά. Αποχές απόρριψη 410 υπέρ. Κατά. Αποχές απόρριψη 411 υπέρ. Κατά. Αποχές απόρριψη 412 και 13 ταυτίζονται υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4-14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4-15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.17 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Δεν ναι, είναι σαφές. Πάμε λοιπόν. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 4.17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει αμέσω. «37 υπέρ 18 κατά». Τώρα είναι σαφές. Τώρα είναι σαφές. Ε, δεύτερο τμήμα υπέρ Αποχές απορρίπτεται. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 420 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 424 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 425 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 426 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 427 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 το δεύτερο τμήμα μόνο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 429 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 430 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 4.31 υπέρ. Κατά Αποχέ απορρίπτεται. 432 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίθηκε. Η 4.33 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Η 4.34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 435 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 437 υπέρ. Και την 36 την κάνατε. Ωραία, συγγνώμη, 436 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα η 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 438 υπέρ. κατά. Είχα πει υπέρ. Υπέρ ξανά. Κατά. Αποχές. Α, τώρα κατάλαβα. Μάλλον απορρίπτεται. 439. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 440 έχει αποσυρθεί. 441 Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4,42 και 43 μαζί Είπε. Κατά αποχές εγκρίνονται. 4,44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4.45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.48 χωριστή, μάλλον κατά τμήματα ψηφοφορία, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Εξίσου εγκρίνεται. 4,49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4,50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4,51. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4,52 υπέρ. Από, υπέρ αποχές εγκρίνεται. 4,53 πρέπει να κάνουμε κατά τμήμα ε, ψηφοφορία, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Α, καταπίπτει. Πάμε στο τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.54 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξω όχι 4.57 4,57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Check. 457, we're checking on... Ηλεκτρονικός έλεγχος στις 4.57. Άρχεται η ψηφοφορία. 4.57 είπαμε. Α, όχι, 458 λέει τώρα ο πρόεδρος. 458. 458. Λοιπόν, ακυρώνουμε λέει ο πρόεδρος. Τι ψηφίζουμε. Την 457. Την 457 λέει ο πρόεδρος. Και έχουμε έναν ε, του ΕΛΚ παραπάνω. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 457 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ ψήφισα λάθος, νομίζοντας ότι ψηφίζουμε την επόμενη. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία ξανά τις 4.57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και τώρα την 4.58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4,59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εντολογικές σκέψεις. Ε, υπέρ το 4 κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ συμβαστική ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Favor. Against. Abstentions rejected. 4. Favor. Against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 το illegal παράνομα να το κάνει illegally. Παρανόμος. Το παράνομα να γίνει παρανόμος. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την 26 η προφορική τοπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 και 29 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά απο... για να ελέγξω ηλεκτρονικά παρακαλώ ε, συμβαστική 30 ηλεκτρονική ψηφοφορία Ακόμα και στη συμβαστική δεν είδα να σηκώνονται χέρια. Λοιπόν, άρχισε και τελείωσε η ψηφοφορία. 53 υπέρ 4 κατά. <laughs> Παρακαλώ, ψηκώστε τα χέρια σας. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 και 41 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 40 και 42 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 και 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 51 το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Εγκρίνεται. 56. 55. Απορρίπτεται. Είπα, ναι, λυπάμαι λέει ο πρόεδρος. Είπα κατά λάθος εγκρίνεται. Απορρίφθηκε η 55. 56. 57. Υπέρ. Ένα λεπτό. 56. Την 56 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τώρα ψηφίζουμε σε όλες μαζί unblock μπλόκ την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Γυναικείων Υποθέσεων. Προ, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτονται όλες ομαδικά. Και τώρα ψηφίζουμε νο, όχι. Α, λι... Συγγνώμη, συγγνώμη. Έχουμε ακόμα την Επιτροπή Αναφορών, τη, τη δέσμη των ε, τροπολογιών της Επιτροπής Αναφορών. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται και αυτές. Η Επιτροπή Γυναικών και Αναφορών ε, δεν Τροπολογίες δεν πέρασαν και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ναι, έληξε η ψηφοφορία. 32 υπέρ, 24 ψήφοι κατά, μία αποχή. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Φλασίκοβα Μπενόβα και παρακαλώ μην μας τέτοιο, μην μας ξαναφέρετε τέτοιο λαχείο παρακαλώ ούτε καν να το διανοηθείτε να ξαναπεράσουμε αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ και έχουμε μια Α, τελευταία ψηφοφορία για μια επιστολή ένα σχέδιο γνωμοδότηση μορφή επιστολή, το οποίο πρέπει να το ψηφίσουμε, είναι από τον Πρόεδρο εμένα, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, για την πρόταση ενός κανονισμού του Συμβουλίου για συγκεκριμένες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν την προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θέλω να σας πενθυμίσω ότι χτες υιοθετήθηκε η μερίσια διάταξη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για σήμερα και περιλάβαμε αυτό το νέο σημείο 16β είναι μια επιστολή της κυρίας Μπάουλς, η οποία είναι πρόεδρος της Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής και αφορά ακριβώς τις νέες εξουσίες, τις προτινόμενες εξουσίες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την προληπτική εποπτεία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε όλα τα μέλη έχει σταλεί αυτή η επιστολή και επειδή το θέμα είναι επίγον, διότι η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα γίνει προς τα τέλη Νοεμβρίου, α, 28-29 Νοεμβρίου, πρέπει εμείς να υιοθετήσουμε αυτή την επιστολή σήμερα. Μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ επί της επιστολής. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. και έληξε η ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Τελείωσε. 42 υπέρ, μία ψήφος κατά, τρεις αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και τη σκληρή εργασία. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με το 17. Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια. Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματο και διαχείριση των κρίσεων. Εισηγητή ο συνάδελφός μας, Σαλβατόρ Γιακολίνο. Έχουμε και τις τροπολογίες για την πρόταση κανονισμού. Έχουμε 57 τροπολογίες που προσθέθηκαν στις 32 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης, συνολικά 90 επί της προτάσεως της Κομισιόν. Η ψηφοφορία προσανατολισμού θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας και ας ακούσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνη, μετά την Επιτροπή και τον εκπρόσωπο της Προεδρίας και τυχόν μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ο συγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το οικονομικό αυτό εργαλείο θα μας βοηθήσει ε, για να εξασφαλίσουμε μονοδοτική στήριξη της αστυνομική συνεργασίας, τη πρόληψη, και καταστολή εγκληματικότητα και τη διαχείριση των κρίσεων. Έχουμε 90 ε, τροπολογίες. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις ε, οι οποίες ε, ακούστηκαν μέσω συγκεκριμένων και σοβαρών προτάσεων, πολύτιμες συνεισφορές από πλευράς των συναδέλφων. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη κύριε Γιακολίνο. Κοιτάξτε, λίγο ησυχία, συνάδελφοι. Σας ζητώ σας ζητώ ε, πολύ ευγενικά να μην μιλάτε για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον κύριο Γιακολίνο. Κύριε Έγγελε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γιακολίνο. Όπως σας έλεγα, υπάρχουν ε, και κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις, οι οποίες διερευνώνται αυτή τη στιγμή και θα συμφωνηθούν τις επόμενες μέρες με κάποιους από τους συναδέλφους και θα κάνουμε και μία συνάντηση των σκιωδών ε, την επόμενη βδομάδα. Έχουμε προβλέψει έναν διαφορετικά ορισμό για, την, για το οργανωμένο έγκλημα, για την κρίσιμη δομή για επίσης μια άλλη κλίμακα για να ελέγξουμε τους στόχους που πρέπει να επιδεθούν μια νέα κατανομή των πόρων, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο και ευελιξία από πλευρά των εθνικών κυβερνήσεων, νέα κριτήρια και ε, διαγράψαμε και την αναφορά στην, στο κρίση. Ο φάκελος τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή προφανώς ε, έχει σοβαρό αντίκτυπο, σοβαρές συνέπειες και αυτό ούτως ή άλλως το ανέφερε και το υπογράμμισε και ο συνάδελφος Μαρινέσκου. Θα πρέπει εδώ να πούμε επίσης ότι έχουμε προβλέψει και ένα ποσοστό των πόρων που συνδέονται που αφορούν μάλλον κυρίως τις συνοριακές χώρες, τις παραμεθόριες χώρες, αυτό το ποσοστό θα πρέπει να δοθεί σε αυτές τις χώρες, διότι μιλάμε για χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Άρα υπάρχει και δυνατότητα transit, ε, όχι μόνο μετανάστευσης, αλλά και άλλων ε, δραστηριοτήτων. Έχει προχωρήσει, όπως σας είπα, το θέμα, το εξετάζουμε. Και εδώ όμως ε, θα είναι χρήσιμες και πολύτιμες οι συνεισφορές ε, και οι προσφογές από την Κομισιό, το Συμβούλιο και από τους συναδέλφους που θα ήθελαν να παρεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, ο κύριο Γιακολίνο, η Κομισιό. Ίσως ε, η Γενική Διεύθυνση η κυρία Πάικ θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καταρχάς πιστεύω ότι ο εισηγητής αναφέρεται και σε κάποιες, αναφέρθηκε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, άρα δεν θα μπορέσω να σχολιάσω. Ε, θα ήθελα όμως να κάνω κάποια πιο γενικά σχόλια για τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και από, την, ε, από τα μέλη σας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια και άλλες προτάσεις για μέσα χρηματοδοτική στήριξης που έχει υποβάλει η Κομισιό για τα εσωτερικά θέματα. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια σχόλια τα οποία εν συντομία, τα οποία είχα έχω επαναλάβει, καταρχάς στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οπου για τον οποίο έχουν υποληθεί πολλές τροπολογίες, η Κομισιό δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε δράση ε, χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα σέβεται τις ε, κοινοτικέ και τις διεθνείς νομοθεσίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, προφανώς. Και ε, έχουμε φροντίσει το κείμενο να το καθιστά αυτό σαφές και μέσω των εκτιμώντας. Αλλά ίσως και αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να εξακριβώσουμε κατά πόσον υπάρχει και να εξασφαλίσουμε και μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς. Όπως είπα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις επίσης, η Κομισιό ε, συνειδητοποιεί ότι οι αρχικοί δείκτες ε, οι οποίοι είχαν υποβληθεί στην πρώτη πρόταση χρήζουν περαιτέρω συζητήσεων. Και σαν αποτέλεσμα αυτού είχαμε κάποια σεμινάρια και κάποια workshops όπου συμμετείχαν τα κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καθορίσουμε τους κατάλληλους κοινού δείκτες. Αυτοί οι δείκτες ε, είναι γνωστοί στην Προεδρία και έχουν διαβιβαστεί από την Προεδρία στην Επιτροπή σας. Επομένως αυτό είναι κάτι παραπάνω από το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Δεύτερον, η εξωτερική πτυχή. Καταρχάς, ε, έγινε μια πρόταση να διαγραφεί η αναφορά στην εξωτερική διάσταση. για το μέσο χρηματοδοτικής στήριξη στην αστυνομική συνεργασία. Και αυτό αναφέρεται και σε ένα ενημερωτικό δελτίο, γιατί εμεί πιστεύουμε ότι το μέσο αυτό θα έχει, πρέπει να έχει περιορισμένη δυνατότητα να παρέμβει σε σχέση και σε τρίτες χώρες. Επίσης, πάλι για την εξωτερική διάσταση υπάρχουν τροπολογίε που προτείνουν να συμπεριλάβουμε στο κείμενο και έναν μηχανισμό συντονισμού. Δηλαδή, ανάμεσα στις, ε, ε, στις υπηρεσίες εξωτερικής συνεργασίας της Κομισιόν και σε άλλους φορείς. Όπως σας είχαμε πει τότε και τον Οκτώβρη, πιστεύουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, καταρχάς. Δεύτερον, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε επαρκή συντονισμό και με άλλα ε, κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, όχι μόνο στην εξωτερική διάσταση αλλά και στην εσωτερική διάσταση. Και πιστεύουμε ότι ο κανονισμός δεν αφορά μόνο τον κανονισμό, δεν πρέπει να αφορά τον κανονισμό θα μπορούσαμε όμως να προτείνουμε στο εκτιμώντας 25 που αναφέρεται στην συνοχή των μέσων που χρηματοδοτώνται μέσω αυτού του μέσου, ε, ένα κείμενο το οποίο να λέει ότι για να εξασφαλίσουμε αυτή την συνοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης θα χρησιμοποιήσει πλήρως τους υπάρχοντες μηχανισμούς συντονισμού και θα τους ενισχύσει ή δυνατόν ή, ή αν παραστεί ανάγκη. Υπάρχουν επίσης πολλές τροπολογίες που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπόλ. Ε, εμείς ε, προφανώς ε, εκτιμούμε το έργο της Ευρωπόλ, όπως και των άλλων κοινοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της, πολιτικής, της εσωτερικής μας πολιτικής και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την εργασία της Ευρωπόλ. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κείμενο και σας υπενθυμίζω ότι η δυνατότητα για τις νομοθετικές αρχές να καθορίσουν ε, περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπόλ θα έρθει όταν η Κομισιόν υποβάλει την πρόταση για τον κανονισμό για τη νέα νομική βάση της Europol. Εν κατακλείδη, να αναφερθώ σε τροπολογίες ε, που ίσως να προέρχονται από κάποιες παρανοήσεις. Η 31 αναφέρεται στην διαγραφή οποιασδήποτε αναφορά στις ιδιωτικού, ιδιωτικές και δημόσιες συνεργασίες. Ε, και πώς δικαιολογείται αυτή η τροπολογία, ότι υπάρχει ένας φόβος ότι ε, είναι σαν να προωθούμε μια ιδιωτικοποίηση της δημόσιας τάξης, της διαφύλαξης δημόσιας τάξης. Προς Θεού δεν τέτοια πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας όταν συζητάμε για συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι να εμπλουτίσουμε τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το δημόσιο για να ε, προωθήσει την ε, δημόσια τάξη. Και εκεί που δεν μπορεί από μόνο το δημόσιο να μπορεί να ε, συνεργάζεται και με το ιδιωτικό τομέα. Η Κυπριακή Προεδρία, η κυρία Χατζικονόμου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώς η συνάδελφός μου κολλείεται σήμερα λόγω έκτακτη ε, έκτακτης αλλαγής της πτήσης, αλλά θα εκπροσωπήσω εγώ την Προεδρία. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για ε, την ευκαιρία που δίνετε στην Προεδρία να λαμβάνει το λόγο για αυτό το θέμα. Η ομάδα εργασίας ad hoc του Συμβουλίου ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών της στις 15 Οκτωβρίου με τις διαπραγματεύσεις τώρα να έχουν μετατεθεί στο, του, στο επίπεδο του Συμβουλίου. 5 Νοεμβρίου, εχθέ, δηλαδή, έγινε η πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου. Είχαμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε μια σειρά ζητημάτων. Η Προεδρία έχει την πρόθεση να μεταφέρει τα δύο θέματα στο Κορεπέ, Τι εννοώ, το ISF για την αστυνομική συνεργασία και το ISF για ε, τα σύνορα και τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Μέχρι τις 15 του μηνός λοιπόν προτιθέμεθα ε, και συγκεκριμένα στις 15 να το φέρουμε στο Κορεπέρ για να πάρουμε εντολή και να αρχίσουμε τις ε, επίσημες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στόχος της Προεδρίας είναι να γεφυρώσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο στο βαθμό του δυνατού πριν τις 19 Δεκεμβρίου που θα είναι η τελευταία συνεδρίαση του Κορεπέρ για την Κυπριακή Προεδρία. Υπό την έννοια αυτή και αφού έχω το λόγο θα ήθελα να διατρανώσω και πάλι εξ ονόματος της Προεδρίας την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε στενά όσο και εντατικά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξουμε σε ε, συμφωνία το συντομότερο δυνατό για τα σχετικά θέματα. Και ένα τελευταίο που είναι εξίσου σημαντικό θα θέλαμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε για την πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Είδα και ένα χέρι να σηκώνεται της κυρίας Αρχεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια στιγμή να βάλετε τα ακουστικά σα Γιατί έχω τι τροπολογίε μπροστά μου στα ε, Ολλανδικά. Οπότε για αλλαγή να μιλήσω Ολλανδικά που δεν το συνηθίζω. Απουσία... Ε, ε τη συναδέλφου Ρόιτοβα θα ήθελα να κάνω εγώ κάποιες ε, προτάσεις. Ε, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για την τροπολογία 61 του κυρίου Ταβάρες ε, για τις ΔΙΤ. Ναι, πραγματικά το έχουμε κάνει αυτό γιατί φοβούμαστε στα θέματα ασφαλείας μιας ΔΙΤ, συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα και τη διατηρούμε την τροπολογία υπαριθμών 61. Και έχουμε και δύο άλλες τροπολογίες των πρασίων που ανέφερε ο εισηγητής στην 75 και την 79 που και οι δύο αφορούν τη χρηματοδότηση μέσων και μέτρων ασφαλείας όπου ε, είναι ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή με τις δικές μας τροπολογίες υπάρχει δυνατότητα να μην χρησιμοποιούνται κοινοτικά κονδύλια ε, για σχέδια όπως είναι το Index και το Clean IT. Τι σχέση έχει αυτό, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείτε ένα τέτοιο πρόγραμμα από κοινοτικά κονδύλια, διότι δεν ε, ευθυγραμμίζονται και συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Γιακολίνο, τι πιστεύει ε, για τις τροπολογίες των Βρασίνων υπαριθμών 75 και 79. Ευχαριστώ. Okay, thank you. If no more... Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους βουλευτές να ζητούν το λόγο. Οπότε, δώσουμε αμέσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο. Παρακαλώ. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Γιακολίνο στην ερώτηση που σα έκανε η κυρία Σαρχεντίνη. Άκουσα και την ε, παρέμβαση της Κομισιόν αλλά και του Συμβουλίου για ένα θέμα το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά, είναι αρκετά όριμο, όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση ε, με τους συναδέλφους μέσω μιας ε, συνάντησης των σκιωδών εισηγητών, όπως είπα και προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία 75 του κυρίου Ταβάρες, όπου ζητάει ο κύριος Ταβάρες μια ψηφοφορία για τον σεβασμό των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Ε, λέγεται στην έκθεση κυρίας Φοντάνα ότι οι προτάσεις που αφορούν το που, ε, προτάσεις χρηματοδότησης Κομισιό πρέπει να, γίνει, να γίνεται μία αξιολόγηση εξάντε Δεν προβλέπεται όμως μία δαπανηρή εκεί ε, διαδικασία. Ο κύριος Σταβάρες βέβαια έχει υποβάλει και άλλες τροπολογίες που έχουν εξεταστεί και θεωρητικά θα γίνουν δεκτές. Ενώ όσον αφορά την τροπολογία με αναφερά στην χρηματοδότηση του μέσου για υποστήριξη στις, για τις τρίτες χώρες. Εδώ η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ανεξάρτητα σε μια πρωτοβουλία της Κομισιόν. Τούτου λεχθέντος επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί και διαθέσιμοι να βρούμε λύσεις καλύτερες και πιο συνεκτικές ε, για αυτό το χρηματοδοτικό μέσο το οποίο έχει σαν στόχο να καταπολεμήσει την, ε, το οργανωμένο έγκλημα. Και εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και θα δημιουργεί έναν μηχανισμό ο οποίος θα συνεργάζεται με τα υπάρχοντα συστήματα. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας είναι αντικείμενο δραστηριοτήτων που εξετάζει συνεχώς η Κομισιό Επομένως θα πρέπει να βρούμε πόρους που αποτελεσματικά θα ενισχύσουν το πρόγραμμα. Το έχουμε κάνει αυτό πρακτικά, δηλαδή δίνουμε περισσότερους πόρους στα εθνικά προγράμματα, διότι πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή κάθε παρέμβαση θα πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται με βάση την τις αποτελεσματικές απαιτήσει, τις ουσιαστικές μάλλον απαιτήσει των κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και μια γενικότερη κοινοτική απέτηση η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Λοιπόν, για την τροπολογία 76 εγώ τροπολογία Ταβάρες έχω κάποια επιφύλαξη και το έχω πει κιόλα αυτό και θα το συζητήσουμε τροπολογία ε, τροπολογία 75. Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχω τη δυνατότητα με τον κύριο Ταβάρες να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ε, και άλλες παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή, σταματάμε εδώ. 27 ε, Νοεμβρίου η προσανατολιστική ψηφοφορία και το, τα θέματα που αφορούν το χρηματοδοτικό μέσο και που... Το, μάλλον το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια και έχει συγκριθεί τον κύριο Μαρινέσκου. Δεν είναι εδώ. Α, εδώ είναι. Α, εδώ είναι. Οπότε συνεχίζουμε με το σημείο 18. Ζητώ συγγνώμη. Δεν σας είχα εντοπίσει θα ζητούσα να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά να και είσαστε εδώ, συνεχίζουμε. Υπάρχει η έκθεση για τα εξωτερικά σύνορα και για τις θεωρήσεις, 180 τροπολογίες. Το λόγο τον έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μαρινέσκου, και μετά από τους εκπροσώπους της Κομισιόν του Συμβουλίου και θα ακούσουμε και κάποιες παρατηρήσεις από τα μέλη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου πρέπει να ε, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσους έχουν υποβάλει ε, τροπολογίες σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Οι τροπολογίες τις οποίες έχω υποβάλει εγώ κυρίως αναφέρονται στον στόχο της εισαγωγής προτύπων για την ασφάλεια των συνόρων και για στην εναρμόνιση όσο το δυνατόν περισσότερο το επίπεδο της ασφάλειας των, ε, των εξωτερικών συνόρων. Και επίσης θα πρέπει να διατεθούν και τα απαραίτητα κονδύλια προς αυτό το σκοπό. Δεν έχω αλλάξει την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων, των κονδυλίων, αλλά προτείνω μια, ένα διαφορετική μέθοδο καταμερισμού. Θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να διατεθούν μετά από την ολοκλήρωση του διαλόγου με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποια μέτρα χρειάζονται ποιες πιστώσεις οι συνάδελφοι μου έχουν υποβάλει πολλές τοπολογίες που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να προτείνω να συμπεριλάβουμε αυτά τα σχόλια στο μέρος εκείνο που αναφέρεται σε αυτή την ουσία Δηλαδή να μην υπάρχει επικάλυψη και να μην επαναλαμβανόμαστε όταν συζητούμε την έκθεση, στην έκθεση αυτή, να μην υπάρχουν επικάλυψη και επαναλήψεις. Ο πρόεδρος ε, απευθύνουμε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, η κυρία Πάικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είχα την δυνατότητα σε προηγούμενη συνεδρίαση να σχολιάσω τις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Θα κάνω και πάλι μερικά σύντομα σχόλια γενικής φύσεως, ε, τα οποία προκύπτουν από τις τροπολογίες που διάβασα. Καταρχά παραλαμβάνω αυτό που είπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σημειώνω τι προθέσει του εισηγητή να, βρει, να βρει την κατάλληλη θέση στον κανονισμό. Έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά από όλε τι δράσει που χρηματοδοτηθούν. Ήδη έχω πει ότι το κείμενο τη Κομισιόν έχει ήδη ξεπεραστεί ω αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχει γίνει με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, ε, καταρχάς, ε, ε, όσον αφορά τη διαγραφή της εξωτερικής πτυχής, πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει καταλάβει ότι χρειάζεται η εξωτερική διάσταση. Τώρα σχετικά με το συντονισμό, με την, σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, δεν νομίζω ότι είναι σωστό σε αυτό τον κανονισμό να αναφερθεί ο μηχανισμός, αλλά στα εκτιμώντας θα μπορούσε να γίνει αυτή η αναφορά. Μετά μάλιστα από το εκτιμώντας 25, Πιστεύω ότι ορισμένοι προσπα... Ε, επισημούν να αναγραφεί πράξεις κατ' εξουσιοδότηση αντί για πράξεις προς Αντί για εκτελεστικές πράξεις. Εγώ προτιμώ την κοινή συνεννόηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μία, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σέβεται αυτή την κοινή συμφωνία και δεν θα χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη αρμοστό είτε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση είτε τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, εν συνεχεία, όσον αφορά την βοήθεια σε περίοδο ή σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, ε, δεν αναγράφεται, δεν περιλαμβάνεται και αυτό το βρίσκουμε ιδιαίτερα λυπηρό, ιδίω στι σημερινέ περιστάσει κρίση. Είχαμε πει ότι θα διαθέσουμε ένα κονδύλι, ειδικά για εξαιρετικέ περιστάσει. και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή σα να διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα υποστή... υποστήριξη σε περιστάσεις εκτακτής ανάγκη. Επίση βλέπω ότι Um, ότι έχει διαγραφεί η αναφορά την οποία ήθελε το Συμβούλιο ε, για τα έξυπνα σύνορα, smart borders, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η αναφορά να διατηρηθεί. Βεβαίω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν εάν στο μέλλον θα διατηρηθεί ή θα υπάρξει ένα σύστημα έξυπνων συνόρων, smart borders, αλλά δεν είναι εδώ ακριβώς ε, η κατάλληλη, το κατάλληλο σημείο να αποτελειώσουμε αυτή την ιδέα. Ως τώρα, σχετικά με το στόχο των ε, κονδυλίων αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια σύγχυση. Υπάρχουν τροπολογίες και από τα μέλη αλλά και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που προτείνουν να συμπεριληφθεί επίσης και το άσυλο. Στο πεδίο εφαρμογής αναφέρουμε ε, του κανονισμού. Προσέξτε λοιπόν, μήπως υπάρχει κάποια επικάλυψη με το Ταμείο Μετανάστευσης ε, στην απόφαση περί κονδυλίων και επίσης οι τροπολογίες που αφορούν τη Frontex την υπηρεσία Frontex, όπως και με την Europol, ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα το ρόλο της υπηρεσίας στη συνεργασία με την Κομισιόν και αναφορικά με την υλοποίηση της πολιτικής εσωτερικών υποθέσεων. υπάρχουν αρκετές τροπολογίες ε, μελών που αντιφάσκουν, ε, πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ορισμένοι θέλουν τη διεύρυνση ε, των αρμοδιοτήτων της ε, Frontex πέραν του σημερινού της ρόλου. Παραδείγματος χάρη στην τροπολογία 55 να υπάρξει ένας κατάλογος προτεραιοτήτων. Ε, και στο, στην τροπολογία 207. Σας είπα ότι εμείς ε, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υποστήριξη της Frontex και ε, ε βάσει του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλειας θέλουμε ασφαλώς να χρησιμοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο και πλήρως όλα τα κονδύλια για τις δράσεις που αναπτύσσει η Frontex. Και γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις δράσεις υπόψη μας, τις οποίες θα αναφέρουμε του χρόνου όταν θα προετοιμάζουμε τα ετήσια προγράμματα των κρατών μελών. Γι' αυτό θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα τα πρότυπα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά τη λειτουργία της Frontex. Από την άλλη πλευρά, στο εκτιμώντας 12, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πρόταση να διαγραφεί συμπληρωματικότητα μεταξύ των κονδυλίων της Frontex και των κονδυλίων αυτού του μέσου. Δεν καταλαβαίνω γιατί επισημείται αυτή τη διαγραφή. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Η Frontex έχει ένα περιορισμένο προπολογισμό και θέλουμε να ξέρουμε ότι μπορεί να εστιάσει η Frontex σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και εν συνεχεία υπάρχει το συμπληρωματικό σκέλος ε, από τα κράτη-μέλη για τις συμπληρωματικές ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει μεταξύ Frontex και κρατών μελών το συμπληρωματικό στοιχείο για την καλύτερη δυνατόν διαχείριση των δράσεων. Αυτά είναι τα σχόλια που θέλω να κάνω. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Κομισιόν, τώρα από πλευράς Κυπριακής ε, Πρόεδρης, κυρία Αργυροπούλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, όπως σας είπα και πριν. Επαναλαμβάνω ότι θέλουμε το θέμα αυτό να συζητηθεί στην Κορεπέ 15 Νοεμβρίου, όπου πιστεύουμε να μας δοθεί η εντολή για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τον επίσημο τριμερή διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο μέλος επιθυμεί να μιλήσει. Καταρχάς, η κυρία Φλότρο που είναι η συγκήτρια ε, της Επιτροπής μας στην, στην ΑΦΕΤ. Ναι, για συντάκτρια γνωμοδότηση είμαι. Η Επιτροπή Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα που ακούσαμε και στις 6 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τη γνωμοδότηση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 36 υπέρ, 6 κατά και 3 αποχές. Ε, εκπλήσουμε πολύ από αυτά που μας λέει για το άσυλο η Κομισιόν, γιατί ακριβώς το άσυλο και η μετανάστευση και το αντίστοιχο ταμείο δεν μιλάει για σύνορα. Οπότε θεωρούμε απολύτως απαραίτητο να μπει ε, στο παρόν χρηματοδοτικό μέσο το άσυλο για τα σύνορα, έτσι ώστε ακριβώς εκεί που είναι τόσο ευαίσθητο το σημείο να έχουμε την εγγυημένη την προστασία εκείνων που χρειάζονται και ζητούν διεθνή προστασία και να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης, non refoulement. Αυτή είναι μία ε, δράση και μία επιλογή που υιοθέτησε και η Επιτροπή Εξωτερικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνοχή των κοινοτικών πολιτικών, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών επιμένει στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, έτσι ώστε η διαχείριση των συνόρων να μην είναι ποτέ αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν ε, την εξωτερική μας δράση. βλέπετε άρθρο 21 της συνθήκης. Η γνωμοδότηση επίσης της Επιτροπής Εξωτερικών λέγει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είπε και η Κομισιόν έτσι ώστε σε καμία περίπτωση ε, να μην διακυβεύονται ε, οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε να παραβιάζονται και επίσης θα πρέπει να επιτρέπεται η χρηματοδότηση δυνατοτήτων παρακολούθησης εκ μέρους των κρατών μελών σε στενή συνεργασία και συνάφεια με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σύνορα. Επίσης, η γνωμοδότηση για ένα θέμα πολύ σημαντικό που μπορεί να σας φανεί εσάς απλώς σημειολογικό αλλά είναι πολιτική σημασίας ε, φρόντισε να κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην αρχή της απειλής, την έννοια της απειλής του κινδύνου και της πρόκλησης. Άλλο απειλή λοιπόν, άλλο κίνδυνος, άλλο πρόκληση. Και είναι σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση γιατί το παρόν μέσο καλείται να ευθυγραμμιστεί και σημασιολογικά και σημειολογικά με άλλους κανονισμούς ήδη ε, εγκεκριμένους και υφισταμένους συγκεκριμένους έτσι, σε ό,τι αφορά τη Frontex. Γνωρίζουμε, έχουμε εργαστεί και ε, σχέση με την έννοια του κινδύνου, του ρίσκου, η ανάλυση του κινδύνου, ας πούμε, της Frontex ε, και ε, υιοθετήσαμε αυτή την έννοια του κινδύνου αντί για απειλή και επίσης όπου χρειαζόταν και ήταν αυτό εύστοχο δεν μιλούσαμε για απειλές αλλά για προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, αντικαταστήσαμε τον όρο της διευκόλυνσης ε, των νομίμων ταξιδιών. Αυτό που, που το βρήκατε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην ε, βιβλιογραφία. Εμείς μιλούμε για κινητικότητα, για ε, νόμιμη μετανάστευση και υιοθετούμε όρους που χρησιμοποιούνται σε άλλα κείμενα που ήδη έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο, όπως είναι ε, να οργανώνεται και να διευκολύνεται η νόμιμη μετανάστευση. Αυτό μας φέρεται πιο ακριβές, πιο σοβαρό και κυρίως παραπέμπει σε κείμενα που έχουν ήδη εγκριθεί από την Ένωση. Αυτά λοιπόν και ε, στη συνέχεια ενίσχυση ε, τις σχέσεις ε, της δράσης των θεωρήσεων και της κινητικότητας για να βεβαιωθούμε και να αγγιθούμε ότι στα σύνορα θα είμαστε σε θέση να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις βελτιώνοντας όσο γίνεται τις δυνατότητες του κώδικου για τις προξενικές θεωρήσεις και την προξενική προστασία ε, για να διευκολύνεται η κινητικότητα των προσώπων. Αυτές είναι οι διάφορες πτυχές. Πέντε βασικά σημεία στη γνωμοδότηση και στις τροπολογίες όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την 6η Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και τώρα τα υπόλοιπα μέλη. Η κυρία Κέλλερ ζήτησε πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ε, τον εισηγητή και το συντάκτη της γνωμοδότησης. Τη συντάκτρια ακούσαμε διάφορες ε, απόψεις. Για μας τους πρασίνους ε, σημασία έχει το Ταμείο των Συνόρων να μην ε, προσανατολίζεται μόνο στην ασφάλεια των συνόρων, την εξασφάλιση των συνόρων, δηλαδή το κλείσιμο, αλλά να είναι και η άλλη όψη του νομίσματος να εξασφαλίζει την κινητικότητα, γιατί τα σύνορα είναι για να τα περνάει ο κόσμος, είναι και γι' αυτό και θέλουμε να μπορεί να τα περνάει να διευκολύνεται δηλαδή και η κινητικότητα, όχι μόνο η ασφάλεια εντό των συνόρων. Βεβαίω έχει σημασία για μα το θέμα τη ε, υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να γράφονται όπου πρέπει και όπου χρειάζονται. Γιατί καμιά φορά έχουμε πολύ συγκεκριμένε προτάσει για πολύ συγκεκριμένε παραγράφου και διατάξει και μετά δεν θα έχει τόσο νόημα να μπει σε μια παράγραφο και όχι σε άλλη, γιατί θέλουμε να συνδέεται ακριβώ εκεί που ανήκει. Ε, η εξωτερική διάσταση ακούστηκε. Εμείς διαφωνούμε με τη διάσταση αυτή και προβληματιζόμαστε. Γιατί είναι επιθυμητό αυτό πολιτικά, είναι αναγκαίο, είναι και νόμιμο, άραγε διότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποτίθεται ότι ασχολείται με τα εσωτερικά. Από την άλλη έχουμε την εξωτερική δράση που είναι θέμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και τώρα τα αναμειγνύουμε αυτά τα δύο και παίρνουμε χρήματα από τον ε, προπολογισμό για τα εσωτερικά για να χρηματοδοτούμε εξωτερικές δράσεις. Θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε μελετήσει φαντάζομαι τις νομικές δυνατότητες, τι δυσκολίες έχετε βρει εκεί και πώς μπορούν αυτές να ξεπεραστούν. Πάντως όταν θα ψηφίσουμε θα το κοιτάξουμε και παρακαλώ κοιτάξτε το αν τέτοιο πράγμα θέλουμε. Να πάρουμε λεφτά από τις εσωτερικές δράσεις για να χρηματοδοτήσουμε εξωτερικές, τέτοιο θέμα θέλουμε. Για τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και τα λεγόμενα έξυπνα σύνορα πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτό το μέσον, σε αυτό το ταμείο, να εντάξουμε θέματα και να βρούμε κονδύλια για το Eurosur και τα έξυπνα σύνορα που δεν το έχουμε ακόμα αποφασίσει. Και μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει καν νομοθετική πρόταση. Και έρχεται στο κείμενο για τη χρηματοδότηση. Μα πώς είναι δυνατό αυτό. Δεν, δεν λέω ότι δεν θα περάσει αυτή η πρόταση, αλλά δεν είναι εδώ το σημείο για να γεννηθεί αυτό το θέμα των, των ε, έξυπνων συνόρων. Ακόμα δεν μας έχει απασχολήσει. Τώρα θα βρούμε λεφτά για κάτι που δεν υπάρχει και ε, που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει ποτέ. Θα πρέπει να εξασφαλίζουμε κονδύλια μόνο για ειλημμένες αποφάσεις και όχι προληπτικά για να το πω έτσι. Επίσης θέλουμε να ανάξουμε τον ορισμό της απειλής στον κίνδυνο και να μιλήσουμε στα σύνορα και να μιλήσουμε για κινδύνους. Γιατί δεν θεωρούμε τη μετανάστευση απειλή, ούτε τους ανθρώπους απειλές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά δεν είναι απαραίτητος απειλές αυτά. Και υποστηρίζουμε τους σοσιαλδημοκράτες στην προσπάθειά τους, στην απόπειρα να βάλουν και ζητήματα που συνδέονται περισσότερο με το Σέγγεν και να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης. Και καλό θα ήταν να εξασφαλιστεί αυτό. Ε, ρώτησε και ο εισηγητής ε, ότι μάλιστα κύριε Μαρινέσκο έχετε αποφασίσει για αυτά τα θέματα. Θα ήταν καλό να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, άλλος ομιλητής. Κύριε Γκυγιόμ, πώς πώς θέλω. Πάρα πολύ γρήγορα. Oui. Ε, Απλώς και μόνο να σας πω ότι όπως είπε και η κυρία Φλότουχα δεν συμμερίζομαι το, αυτά που είπε η Κομισιόν για τον αποκλεισμό των ερωτημάτων για τα θέματα του ασύλου. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε σε ορατότητα και σε διαφάνεια ε, εάν τονίσουμε και αυτή την διάσταση του ασύλου και το δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να θίξω εν συντομία, αφορά την ορολογία. Ε, υπάρχουν Είδαμε σε κάποιες ε, ε, εκθέσεις ε, την ανάγκη να αντικαταστήσουμε το illegal από το irregularité, η τούμπαλιν. Και εδώ είναι θέμα ορολογία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κανείς άλλος δεν θέλει να προσθέσει κάτι. Ας επιστρέψουμε στον εισηγητή, τον κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ και του συναδέλφους που εκφράσαν τα σχόλιά τους, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βρούμε ένα συμβιβασμό στην συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ και την Επιτροπή, την Κομισιόν. Υποστηρίζω σχεδόν όλα τα σχόλια που έκανα η Κομισιόν. Και ευχαριστώ και το Συμβούλιο για την πρόθεση του να οριστικοποίηση και ε, στην και να αρχίσει ο τριμερής διάλογος. Ευχαριστώ πολύ. I'm having problem with my mic, I see. So. Ε, έχω κάποια μικρά προβλήματα με το μικρόφωνο. Λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο. Και για το επόμενο σημείο θα πρέπει να περιμένουμε την εισηγήτρια και γι' αυτό που να έρθει ας κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. So, we thank you because Mrs. McIntyre was the rapporteur in charge. Ευχαριστώ. Και τώρα το επόμενο μας θέμα είναι το πρόγραμμα Περικλής. Η συγγήτρια μπήκε μόλις στην αίθουσα, της δώσουμε ένα λεπτάκι. And get ready to get going. να ετοιμαστεί. Θα ήθελα όμως να πω ότι το σημείο αυτό, το 19, που αφορά ακριβώς τη τη θέσπιση προγράμματο ανταλλαγό εμεί και κατάρτιση για την προστασία του ευρώ, το λεγόμενο περικλή 2020. Ε, στόχος μας είναι σήμερα να εξετάσουμε τις τροπολογίες για το πρόγραμμα αυτό κατάρτισης συνδρομής και ανταλλαγών. 23 τροπολογίες και ε, μαζί με το σχέδιο έκθεση συνολικά έχουμε 42. Ας ε, να σας πω ότι στις 27 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία προς ανατολισμού. Η κυρία Μάκιντάιρ έχει το λόγο, μετά ένα λεπτό η Κομισιόν και το Συμβούλιο και τα μέλη μας. Η κυρία Μάκιντάιρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ που με περιμένατε δεν έχω ακόμα καταφέρει να βρω ένα μαγικό τρόπο να βρίσκομαι σε δύο σημεία ταυτόχρονα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις, τους κοιόδης εισηγητές για αυτή την επ' αυτής της έκθεσης και ιδιαίτερα τη γραμματεία για όλη την υποστήριξη την οποία μας προσέφερε. Και όσοι από σας ε, δεν έχουν πολύ στενή σχέση με το θέμα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα για την ε, συνδρομή στην κατάρτιση πρόγραμματων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κυβδηλία. Δεν είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα και βασικά συμφωνούμε από αυτού. Υπάρχουν ε, ορισμένες τοπολογίες τις οποίες έχω δεχτεί. Είχαμε μία συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών και έχω υποβάλει, έχω συντάξει ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες ε, που έχουν λάβει υπόψη πολλές από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και ε, επίσης ευχαριστώ και την Επιτροπή για όλη τη δουλειά που έκαναν για να μας εξηγήσουν λεπτομερώς τι επιδιώκουν. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών των ενεργειών και με την υποστήριξη ε, ένα-δύο σχεδόν εισηγητών έχω αποσύρει ορισμένε τροπολογίες μου και έτσι υπάρχουν ε, λιγότερες τροπολογίες. Έχει μειωθεί ο τους. Έχουμε δύο επίμαχα θέματα και θα ήθελα πραγματικά να αμβληθεί αυτή η ένταση που υπάρχει μεταξύ τους. Το πρώτο αφορά της πράξεις εξουσιοδότηση Είναι ένας τομέας αυτός που είναι είτε αρμοδιότητα του, της Προεδρίας είτε των, των Προέδρων των Επιτροπών ότι θα πρέπει να υπάρχουν πράξεις κάτω εξουσιοδότηση να αναφερθούν. Και αν δεν υπάρχουν αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση, η έκθεση αυτή θα, δεν θα προχωρήσει στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν έχω περιλάβει μια πρόταση για πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Όμως, σημείωσα ότι σκιώδεις εισηγητές και ιδιαίτερα ο κύριος Διαστημίρα προτείνει να μην συμπεριλάβουμε τις πράξεις αυτές. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή αν τις χρειαζόμαστε στο τελικό κείμενο της πράξης κατά εξουσιοδότηση ή όχι. Το δεύτερο επίμαχο θέμα όπου υπάρχουν διαφωνίες είναι η συγχρηματοδότηση, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Εγώ προτείνω μία δέσμη ε, ποσοστό, μία δέσμη αριθμών και ο στόχος μου ήταν να, καταμεριστούν, να επιμεριστούν σωστά, δίκαια και όσο το δυνατόν πιο ευρέως τα υπάρχοντα λίγα κονδύλια. Ενώ άλλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλότερη συγχρηματοδότηση, υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότηση. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα δύο επίμαχα ε, θέματα, πράξη κατοξιδότηση και συγχρηματοδότηση. Ε, εκτός αυτών συμφωνούμε στα υπόλοιπα και όπως σας είπα μπόρεσε να ενσωματώσω πολλές προτάσεις τροπολογιών στο κείμενό μου. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψη και των άλλων μελών από αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Α, είμαι πρόσωπος της ε, ε η οποία είναι σήμερα υπεύθυνη για το πρόγραμμα Περικλής 2020. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είχαμε μια τόσο καλή συνεργασία με την συγγύητα, την κυρία Μάρκιντάιρ, και χαίρομαι ιδιαίτερα που υποστηρίζει τη συνέχιση αυτού του προγράμματος Περικλής μέχρι, το επόμενο, μέχρι την επόμενη γενιά ε, των δημοσιονομικών προοπτικών έχουν Α, έχουμε αποσύρει την πρόταση να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στα προγράμματα κατάρτισης εισαγγελής και δικαστική εκπρόσωποι. Ε, στη συγχρηματοδότηση όντως υπάρχει ακόμα μια διαφορετική προσέγγιση. Κάνουμε μια μελέτη επιπτώσεων η οποία συνόδευσε την πρότασή μας, το σχέδιο κανονισμού και αυτή η μελέτη επιπτώσεων η οποία έγινε σε συνεργασία με διάφορα σεμινάρια που οργανώθηκαν με ενδιαφερόμενους δικαιούχους από τα κράτη-μέλη και τα λοιπά, αρμόδιες αρχές, τόνισαν το μεγάλο όφελος που προκύπτει από το πρόγραμμα Περικλής και πόσο αποτελεσματικό είναι για την καταπολέμηση της παραχάραξης Είπαν λοιπόν όλοι αυτοί οι κύκλοι ότι θα ήθελα να δουν την αύξηση της χρηματοδότησης. Γενικά πιστεύουμε ότι το 80% δικαιολογείται. Το 80% για χρηματοδότηση δικαιολογείται. Αυτό λοιπόν το ποσοστό αυτή η πρόταση βασίζεται σε όλες τις μελέτες, έρευνες και συζητήσεις που κάνουμε και πιστεύω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Γι' αυτό εμείς εμένουμε στην αρχική μας πρόταση. 80% ε, και 90% για εξαιρετικέ περιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα το επίμαχο θέμα των πράξεων κατευθυνσιοδότηση, ξέρουμε ότι αυτό προέρχεται από τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου και της Προεδρίας. Εμείς, τονίζω, δεν έχουμε υποβάλει καμία πρόταση από αυτού. Διότι, εάν κάναμε μια τέτοια πρόταση, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η υλοποίησή της από την Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη, να εδραιώσουμε, μια, να θεσπίσουμε μια ολόκληρη διαδικασία πράξεων κάτω εξουσιοδότης για τα ετήσια προγράμματά μας. Εάν κάνουμε την εισαγωγή μιας τέτοιας πρότασης, θα είχαμε τουλάχιστον μια δίμηνη καθυστέρηση και διοικητικό άχθος. Θα είχαμε και μεγάλες ε, σημαντικές καθυστερήσεις στη δημοσίευση του προγράμματος. Γι' αυτό δεν θέλουμε να ε, ακολουθηθεί αυτή η κατεύθυνση. Τονίζουμε ότι δεν επισημούμε αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό υποστηρίζουμε την τροπολογία αυτή για τις πράξεις κατεξουσιοδότησης που αφορά τις πράξεις κατεξουσιοδότης. Έχουμε επίσης κατα... δει ότι νομίζω στην τροπολογία 30 θα πρέπει οι δράσεις αυτές να αναφέρονται μόνο στις ανταλλαγές τελεχών δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό ήδη διοργανώνει και έχει καλύψει πάρα πολλά σεμινάρια, εργαστήρια κλπ. Άρα θα πρέπει η υλοποίηση του προγράμματος και οι στόχοι του προγράμματος ε, ήδη εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό και τώρα να εφαρμοστούν αυτά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα μόνο στην ανταλλαγή στελεχών και γι' αυτό δεν υποστηρίζουμε αυτή την τροπολογία. Όσον αφορά το θέμα του, του κοινού, αυτό ήδη το έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει ήδη διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Πιστεύω ότι αυτή την πράξη, αυτή τη δράση θα πρέπει να τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και για το κείμενο για τα πρότυπα της Όλαφ και την Α, είναι οι τροπολογίες 40 και 41 που αφορούν αυτές τις ρήτρες, τις ρήτρες ε, οι οποίες έχουν προταθεί από την συγκήτρια και ε, τις οποίες υποστηρίζουμε θερμά. Ε, υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει από πλευράς Κυπριακής Προεδρίας. Όχι. Ωραία. Δίνω το λόγο στα μέλη. Ο κύριος Δίας Δεμέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια φυσικά είναι λόγια ευγνωμοσύνης και ευχαριστίων προς την κυρία Μάκενταρ. Πάντα είναι πολύ αποτελεσματική στο έργο της. Αλλά θέλω να την ευχαριστήσω και για την ευαισθησία που έδειξε δεχόμενη ορισμένε από τις δικές μου οκτώ τροπολογίες ε, προσπάθησε άλλες να ε, τις συμβιβάσει και βεβαίως σε κάποιες άλλες διαφωνεί. Γιατί και η διαφωνία ε, και η απόκληση είναι και η υγιής πρακτική αλλά και συνήθι στο κοινοβούλιο. Σε δύο τροπολογίες που εγώ όμως θεωρώ εκ των ουκ άνευ και ουσιαστικότατες. Σε αυτές τις δύο τροπολογίες, κυρία εισηγήτρια και κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση και να σας εξηγήσω γιατί. Διότι έχω ευρύτατη εμπειρία στην προστασία του ευρώ. Μεγάλη και κοινοβουλευτική εμπειρία. Και με μια άλλη συμπροματική έκθεση αυτής που είμαι εγώ εισηγητής, έρχονται να συμπληρωθούν 8, 7, 9 εκθέσεις που έκανα εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο και πάντα, πάντα με κριτήριο την προστασία, περισσότερη και την καλύτερη προστασία για το νόμισμά μας. Ε, δηλώνω και δέχομαι ότι είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένο το νόμισμα από τον επαγγελματικό ζήλο της Όλαφ Κυρίως η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το πρόγραμμα Περικλήσεις προστατεύεται και με τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Και μάλιστα σε ελάχιστο κόστος, έτσι ελάχιστο είναι το κόστος, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αυτό είναι το ποσό. Για όλο τον προϋπολογισμό. Και με ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο καταφέρνουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η επίθεση και η παραχάραξη του ευρώ. Είναι πιο ισχυρό το νόμισμά μας και πιο δύσκολο να παραχαραχθεί από το δολάριο, που ξέρετε τι ζωή έχει και πόσα έτη το δολάριο. στη συνέχεια, ε, λέω στην εισηγήτρια μετά από αυτή την εισαγωγή ότι ε, θεωρώ ότι στο ποσοστό ε, χρηματοδότησης είμαι πρόθυμος ε, στις ε, κανονικές περιστάσεις να έχουμε 80% και σε έκτακτες 90%. Για μένα αυτό είναι πραγματικά αδιαπραγμάτευτο, αλλά δεν το κατεβάζω αυτό από το μυαλό μου. Είναι ε, δεδομένο, λογικό και απολύτως απαραίτητο για να συνεχίσουμε την προστασία που τόσο χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια θα ήθελα να πω το εξής. Μήνες, όπως γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι ολόκληρους, αφιέρωσα ε, στη συζήτηση ε, για ε, τις κατεξουσιοδότηση πράξης για τον κανονισμό 539 το 2001 που ήμουν εγώ εισηγητής. Αλλά πρόκειται για μια συμφωνία διοργανική που δεν έχει ακόμα οριστεί και τα ξέρει αυτά ο πρόεδρος Λόπες Ακυλάρ. Το θέμα είναι απλό και εύκολο, δηλαδή πώς θα διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης κατάστασης και συμφωνώ με την Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η έκθεση αυτή δεν ε, είναι έκθεση που θα πρέπει να ε, κατατεθούν εδώ οι κατεξιόδηση πράξεις. Είναι καλή η διαχείριση των προγραμμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να μπει στη διαδικασία ε, κάθε χρόνο το πρόγραμμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Γι' αυτό Συμφωνώ ε, και σε αυτό το θέμα, κυρία ε, ε, εισηγήτρια, με την Όλαφ. Και επειδή τους ξέρω και τους εμπιστεύομαι στην Όλαφ, σας λέω ότι δεν χρειάστηκε και συντονισμό. Συμφωνούμε γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά συμπίπτουμε. Ε, διότι αυτά τα ε, υπαγορεύει η κοινή λογική. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τις πλειοψηφίες που εσείς, κυρία εισηγήτρια, ε, συγκεντρώνετε, και πάρα πολύ θέμητα, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλειοψηφία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έχει εμπειρία στο πρόγραμμα Πέρικλης. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διαστεμέρα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει άλλος ε, το λόγο, άλλο μέλος ε, της Επιτροπής μας. Επιστρέφουμε στην εισηγήτρια την κυρία Μάκιντάιρ για να απαντήσει αν θέλει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και στην την Κομισιό και τον ε, κύριο Δίας Δεμέρα για τα σχόλιά τους. Θα ήθελα απλώς να απαντήσω στην Κομισιό ότι οι δύο συγκεκριμένες τροπολογίες οι οποίες δεν σας ικανοποιούν, που είναι η τροπολογία 30 και η άλλη νομίζω είναι 27, αν δεν κάνω λάθος, και κατά την άποψή μου θα, τους, θα τις απέριπτα κι εγώ, ούτως ή άλλως. Υπάρχει όμως κι άλλη μία που πιστεύω θα πρέπει να απορρίψουμε δεν μπορώ να τη βρω τώρα τέλος πάντων, αλλά ήταν στην, ε, από τις πρώτες τροπολογίες που πιστεύω ότι όντως δεν ταιριάζει στην έκθεση αυτή. Είναι η τροπολογία 20. Επομένως, αυτό το που ήθελα να πω είναι ότι συμφωνώ με την Κομισιό για τις απόψεις της επί των ε, ε, τροπολογιών. Τώρα, για αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις εγώ άκουσα τις συμβουλές που μου δόθηκαν με βάση όσα αποφάσισε η Επιτροπή των ε, Προέδρων των Προσωπιών. Και θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μία άποψη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε αυτές τις ε, της πράξης ε, της κατεξουσιοδότηση, διότι αλλιώς δεν έχω καμία αντίρρηση να δεχτώ αυτό που είπε ο κ. Δίας και να αποσύρω τις τροπολογίες. Εάν, τώρα δεν ξέρω, εσείς θα μπορούσατε πρόεδρε να μας πείτε, γιατί εγώ νομίζω ότι η συνέλευση των προέδρων ε, αυτό αποφάσισε. Ένα πράγμα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα είναι το ποσοστό χρηματοδότηση. Η κατά μου, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και περικοπές. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε να τους σώσουμε μέσω αυτού του προγράμματος, ε, αυξάνοντας τα ποσοστά συγχρηματοδότηση απλώς και μόνο για να αντιμετωπίσουν τις περικοπές τους. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι συμφωνούμε. αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε τον ε, Πρόεδρο κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε αν υπόψη μας ε, τις ε, κατεξουδότηση πράξης. Αυτό το κάναμε, το έχουμε κάνει και με πολύ πιο ειρηνικό τρόπο από ό,τι άλλες επιτροπές που μπλεχτήκανε σε αυτές τις θεσμικές συζητήσεις για, τις, για τα διάφορα είδη των πράξεων. Δεν χρειάζεται κι εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι για να γίνει δεκτή η πρότασή σας θα πρέπει να το συζητήσουμε διμερώς. Γιατί έχει τεχνικές πτυχές αυτό το θέμα και δεν μπορούμε να το λύσουμε επί του παρόντος. Ας τα αφήσουμε έτσι όπως είναι τώρα και προτείνω να, να το συζητήσουμε περαιτέρω για να δούμε ποιο ακριβώς είναι το εύρος, αν θέλετε, της πρότασης που υπάρχει. Και να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το θέμα γραπτά. Επομένως, εάν δεν θέλει κανείς να προσθέσει οτιδήποτε τώρα, δεν θα γίνει καμία άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Α, βλέπω ένα χέρι, βλέπω να ε, δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μάκιντάιρ, την εισηγήτρια, γιατί δέχτηκε και εκείνη συμφωνεί μάλλον να απορριφθούν οι, προτα... οι τροπολογίες 20, 27 και 30. Υπάρχει όμως και άλλη μια τροπολογία την οποία θα έπρεπε να σας την πω, γιατί και αυτή είναι κάπως προβληματική για την Κομισιό, που είναι η τροπολογία 7, η οποία αποκλεί από την κατάρτιση και από το πρόγραμμα Περικλής οι ομάδες εμπειρογνωμόνων. Έχουμε πολλούς... Ε, ε, Πολλέ πολλές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, όπου συμμετέχουν, ε, έχουμε εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές ε, που ακριβώς ε, ευαισθητοποιούν τους, τις αρμόδιες ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες, για το πώς μπορούν να παραχαραχθούν τα, τα νομίσματα. Επομένως, εάν γίνει δεκτή η τροπολογία 7, δεν θα είναι αυτές οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων ε, αντικείμενα κατάρτισης με βάση το πρόγραμμα Περικλής. Επομένως θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Λοιπόν, Εάν δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι, περνάμε στο σημείο 20 που είναι και το τελευταίο για σήμερα. Το θέμα σε ΠΟΛ, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Έχουμε μαζί μας Έχουμε μαζί μας ε, εκπρόσωπο της ΣΥΠΟΛ, τον δόκτορα Φέρεντς Μπάμφι, που είναι ο διευθυντής της έπολου, που είναι έτοιμος να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί με τον κύριο Ράινχαρτ Πρίμπε. Ελάτε εδώ στο βήμα. Κύριε, ο κύριος Πρίμπε ήταν σήμερα το πρωί και στην συνάντηση των συντονιστών. Είναι και εδώ ε, Διευθυντής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Λοιπόν, λάβετε υπόψη σας ε, ότι η Κομισιόν στο τέλος του 2012 και αρχές του 2013 ε, θα υποβάλει μια πρόταση για συναπόφαση έτσι ώστε η, η η πρόταση για την ΣΥΠΟΛ να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, για να προετοιμαστούμε για αυτή την πρόταση, σαν ένα τμήμα, αν θέλετε, της, του της συνεχής ε, συζήτησης που έχουμε, ε, καλέσαμε εδώ τον κύριο Μπάνφη και τον κύριο Πρίμπε για να μας ενημερώσουν για το ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΠΟΛ και ποια θα είναι η αναμενόμενη πρόταση για την ΣΥΠΟΛ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπάνφη και μετά θα αφιερώσουμε και κάποια λεπτά στον κύριο Πρίμπε και μετά τα μέλη της Επιτροπής μας. κυριε μπανφη Μπάμφη, 10-15 λεπτά, όσο θέλετε τέλος πάντων. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕΙ, αγαπητοί συναδελφοί κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι για αυτή τη δυνατότητα που μου δίδεται σαν διευθυντής της υπηρεσίας της, Ακαδημαϊκής, ε, της Αστυνομικής Ακαδημίας να παρουσιάσω εν συντομία τα επιτέχματα της ΕΠΟΛ στην προώθηση της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασίας μέσω του, της μάθησης. Καταρχά να σας περιγράψω τις αλλαγέ που έγιναν από την ΣΕΠΟΛ τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι ε, κυρίω χάρη στην επαγρύπνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ΣΕΠΟΛ μπορεί να ε, πει ε, καθαρά ότι οι επιχειρήσεις της είναι νόμιμες, κανονικές και αξιόπιστες. Από το 2010 τα οι εκκρεμότητε εκκρεμότητες ρυθμίστηκαν. Αυτό έγινε με, με διαδοχικούς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 τις οποίες ε, ε, επιβράβευσε κιόλας ε, για την αποτελεσματικότητά τους το σύστημα προτύπων εσωτερικού ελέγχου. Έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας πιστεύω. Έγιναν αλλαγές οι οποίες είναι μακρόπνοες και αποτελεσματικές σε όλους τους τομείς. Καταρχάς η διακυβέρνηση μπήκε σε κάποια πλαίσια. Οι επιτροπές που συνήθως συνεδρίαζαν τρεις και τέσσερις φορές το χρόνο διαλύθηκαν. Έγινε μια, ένας εξορθολογικός των ομάδων εργασίας της ΕΠΟΛ σύμφωνα με την προσέγγιση ε, result oriented, δηλαδή προσανατολισμένη στον, στο αποτέλεσμα και μία μείωση των συναντήσεων της, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου από 6 σε 2 το χρόνο ε, οδήγησαν σε μία, διαδοχική, σε μία προοδευτική μείωση του, του κόστους από 518.000 ευρώ το 2009 σε 169.000 το 2012. Η... Επίσης επιτεύχθη σημαντική πρόοδος και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο. Ε, οι συνολικές, το συνολικό ποσοστό ε, ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην ΣΕΠΟΛ είναι περίπου στο 93%. Η εκπαίδευση είναι πιο αποτελεσματική. Ο αριθμός των ε, συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της αυξήθηκε από 2.300 το 2009 σε 3.000 σε 4.300 το 2011 και θα είμαστε γύρω στους 5.000 φέτος. Επίσης, ο αριθμός των δραστηριοτήτων από 91 που ήταν το 2010 έφτασε σε 106 το 2011. Ένα από τα βασικά μας προϊόντα, αν θέλετε, είναι το Ευρωπαϊκό ο πρόγραμμα αστυνομικών ανταλλαγών που αυξήθηκε από 50 συμμετέχοντες το 2009 σε 299 το 2011 και καλύπτει 15 θέματα. Ε, καλύπταμε μάλλον 15 θέματα το 2011, τώρα καλύπτουμε 24. Και ε, οι συμμετέχοντες κατά 98,4% αξιολόγησαν το πρόγραμμα καλό ή πολύ καλό. Επίσης ο αριθμός των ε, εικονικών φοιτητών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μέσω του, του ίντερνετ ξεπέρασαν τους ε, φοιτητές που φιλοξενούσαμε και είχαμε 3.016 ε, για τις δραστηριότητες μέσω ίντερνετ και, 100, και, και, συγγνώμη, και 1.497 φοιτητές. Αυτά και πολλά άλλα παραπάνω ε, επιτεύθηκαν με έναν προϋπολογισμό ο οποίος παρέμεινε σχετικά σταθερός 8,5 ε, εκατομμύρια το 2012, 8,300 το 2011 και 7,800 το 2010. Ε, έχουμε 38 άτομα προσωπικό και πέντε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ε, της Ακαδημίας μας. Ε, η προσέγγιση, η εκπαιδευτική μας προσέγγιση έχει ενταχθεί πλήρως στο θεσμικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τους συναδέλφους στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Ε, ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας προέρχεται από, τη νέα, από το νέο κύκλο πολιτικής για το σοβαρό, αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος ή για την υποστήριξη συγκεκριμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως στρατηγική για την, για την ε, εκρίζωση ε, της παράνομης διακίνησης ανθρωπίνων όντων εμείς ε, συνεργαζόμαστε επικοδομητικά και με άλλους ε, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Όμως, αυτό το οποίο δεν βγαίνει από στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται, είναι ο ρόλος της ΕΠΟΛ στην δημιουργία εμπιστοσύνης, εναρμονισμένων πρακτικών και ενθάρρυνσης της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ε, ε, κουλτούρας, αστυνομικής κουλτούρας και αυτός είναι ένας ιστορικός ε, ρόλος της ΣΕΠΟΛ. Η εκπαίδευση της αστυνομίας πρόσφατα και μόνο γίνεται αυτόνομα και αντιμετωπίζεται σαν ένα εργαλείο αστυνομικού επαγγελματισμού. Σε βασική αντίθεση με τον στρατιωτικό κόσμο, οι αστυνομικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν είχαν θεσμοθετημένη εκπαίδευση μέχρι τον προηγούμενο αιώνα τα Ινστιτούτα Αστυνομικής Εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν μετά την δεκαετία του 1960. Πρόσφατα έγινε μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στην πολιτική εκπαίδευση και στην πολιτική κατάρτιση. Η όροι κατάρτιση και εκπαίδευση πολλές φορές χρησιμοποιούνται ε, ο ένας αντί για του άλλου. Όμως διαφέρουν σημαντικά. Η κατάρτιση ορίζεται ε, σαν ε, η παιδεία που έχει σαν στόχο την δημιουργία συγκεκριμένων τεχνικών προσόντων για την ε, ε, εκπλήρωση των πρακτικών καθηκόντων. Η παιδεία όμως αντίθετα ε, στοχεύει στην δημιουργία χαρακτήρα νου και φυσικής ικανότητας του ατόμου. Επομένως είναι κάτι πολύ πιο γενικό. Σε αυτά τα πλαίσια θα αναφερθώ στην πολιτική κατάρτισης της αστυνομίας από μια εκπαιδευτική προοπτική. Σε μια συνολική κοινωνία η αστυνόμευση πρέπει να συνδέεται με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή όπως παρουσιάζεται στην, ε, ε, στην πραγματικότητά μας που ζούμε. Πρέπει να είναι ανοιχτή και σε διάλογο με την κοινωνία. πρέπει να στραφούμε στον διάλογο. Αυτό απαιτεί μια ευρεία γκάμα αρμοδιοτήτων. Η χρησιμοποίηση της φυσικής και της, των, μεθόδων, επιστημονικών μεθόδων και των ερευνητικών μεθόδων στη σύγχρονη αστυνομία και στην κατάρτιση των, την αστυνομική κατάρτιση είναι απαραίτητη. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι η πτυχή εκπαίδευσης θα πρέπει να υπερισχύει σε σχέση με τις άλλες πτυχές. Το κλειδί είναι να βρεθεί το σωστό μείγμα και να αξιολογήσουμε τις συγκεκριμένες αποστολές που πρέπει να υλοποιήσει η παιδεία και η κατάρτιση. Συνειδητοποιώ απόλυτα ότι ζούμε δύσκολους οικονομικούς ε, καιρούς και ε, κάθε ευρώ μετράει. Πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Όμως θα πρέπει να ξεπεράσουμε την απλή λογιστική προσέγγιση. Έχουμε μικρή κλίμακα ε, εξοικονομίας ε, βραχυπρόθεσμες και μικρές, ε, μικρής κλίμακας. Δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα, δεν προσφέρει μάλλον απαραίτητα καλύτερη αποτελεσματικότητα μακροπρόθεσμα. Οι αστυνομικέ υπηρεσίες στην Ευρώπη έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από, την, από τις περικοπές και από την πολιτική λιτότητας. Οι, προϋπολογισμοί έχουν ε, ε, περιοριστεί. Όμως το εργαλείο, αν θέλετε, τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους ε, οι αστυνομικές δυνάμεις στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για τα ποινικά θέματα διευρύνεται. Αλλά δεν χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένο κίνδυνος ότι η γενιά των ε, αστυνομικών αξιωματικών δεν θα έχει μεγάλη πρόσβαση στις δυνατότητες ε, εκπαίδευσης. Όμως, ο βασικός κίνδυνος αφορά τους πολίτες που θα αντιμετωπίσουν μια μείωση στην ποιότητα της αστυνόμευσης. Η όλων θέλει να ενισχύσει την αστυνομική συνεργασία μέσω της παιδείας. Η, η, η κατάρτιση δεν είναι μόνο ε, μια αποκλειστική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αστυνόμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας παράγοντας κλειδί που συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η, Ευρωπαϊκή η ευρωπαϊκή κατάρτιση απαιτεί επενδύσεις και ελπίζω ότι τους επόμενους ε, μήνες θα δοθεί η δυνατότητα ε, να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υποστηρίξει καλύτερη αστυνόμευση μέσω του learning, μέσω της ε, παιδείας. Είμαι σίγουρος ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κατάρτισης θα προσφέρει μια πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. We thank you. We thank you for your... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και προτείνω να ακούσουμε τώρα τον κύριο Πρίμπε. Αν θέλετε και μετά τα μέλη μας. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Στα θέματα εσωτερικής ε, πολιτικής και δικαιοσύνης έχουμε μια σειρά από οργανισμούς και ε, υπηρεσίες. Ε, η ΣΕΠΟΛΗ είναι ένα μικρό μεν μέλος, αλλά πολύ σημαντικό αυτής της οικογένειας που μας βοηθάει να υποστηρίξουμε τις πολιτικές μας και η ΣΕΠΟΛ και το δίκτυό της έχουν ε, διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών στην ε, επιβολή του νόμου. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική ε, και δύσκολη οικονομικά η καιρή και το είπε και το Κοινοβούλιο και το 2010 έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να λυθούν θέματα που εκκρεμούσαν και δεν ε, θέλω να χάσω την ευκαιρία να συγχαρώ το Διευθυντή ε, Πάνφη και το επιτελείο του για την τόσο καλή τους επίδοση και απόδοση τα τελευταία έτη. Ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς υποστηρίζουμε τις ΕΠΟΛ και τις δράσεις της για να φτάσει στους στόχους του προγράμματος της Σοχόλμης για ενίσχυση και περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Και πολλές δράσεις ε, όπως είναι η προώθηση της αστυνομικής συνεργασίας, προγράμματα ανταλλαγών αλλά και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων ε, αποτέλεσαν το πρότυπο και το παράδειγμα για την εκπαίδευση των αστυνομικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άκουσα προσεκτικά τις σοφή διάκριση που κάνατε μεταξύ της παιδείας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης θα μπορούσε ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να βοηθάει και στη διαπαιδαγώγηση ε, των αστυνομικών και να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κουλτούρα αστυνομική, ε, αν κατάλαβα καλά τη διάκριση που κάνατε. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μας εμπνέουν και μας βοηθούν για να ε, δημιουργήσουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπαίδευσης που αυτό τον καιρό καταρτίζεται και στόχο έχει να υπογραμμίσει κυρίως την αστυνομική βεβαίως ε, εκπαίδευση, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα ας πούμε διασυνοριακά, για νέες προκλήσεις, όπως είναι το κυβερνοέγκλημα ή ακόμα και εκεί που καλούμεθα να δώσουμε υποστήριξη σε ε, αποστολές ε, Ευρωπαίων αστυνομικών σε ε, περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε κρίση. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια έχει ανατεθεί στο, στη ΣΕΠΟΛ, στο Διευθυντή και το επιτελείο του. Θα ήθελα όμως επευκαιρία να σας ενημερώσω και για κάποια άλλα θέματα που συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προβληματισμό για τη νέα ε, νομική βάση για τη Europol και τη ΣΕΠΟΛ. Ακόμα είμαστε στο στάδιο των ε, προβληματισμών και της περισυλλογής, τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά όπως ξέρετε και για τις δύο αυτές υπηρεσίες και οργανισμούς θα κάνουμε μέχρι τέλη του έτους προτάσεις για τη νομική βάση και ταυτόχρονα θα παρουσιάσουμε και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπαίδευση. Μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι προτάσει και ένα από του λόγου είναι ότι. Σα είπα, είμαστε ακόμα στο στάδιο ε, του προβληματισμού. Σκεφτόμαστε αν θα έχει νόημα να ε, ε, ενωθούν η ΣΕΠΟΛ με τη Europol να υπάρξει μια συγχώνευση γιατί έχουν κοινή προσέγγιση τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή για τη διαχείριση των κοινοτικών οργανισμών, των agencies. Δηλαδή, κάποιες υπηρεσίε που είναι πάρα πολύ μικρές, μήπως θα ήταν καλύτερο να συγχωνευτούν με κάποιες άλλες. Απλούστατα για λόγους ε, διοικητικών ε, οικονομιών. Δεν έχουμε καταλήξει, το σκεφτόμαστε. Η έκβαση είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν ήθελα όμως να χάσω την ευκαιρία να σας ενημερώσω γι' αυτό. Βεβαίως το γεγονός ότι προβληματιζόμαστε σχετικά δεν σημαίνει ότι αποδίδουμε μικρότερη σημασία στην εκπαίδευση των αστυνομικών μας. Το αντίθετο, μια τέτοια συγχώνευση σε περίπτωση που προταθεί και γίνει κανονικά θα γίνει με κάποιους όρους και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση των αστυνομικών σε μια μεγαλύτερη δομή, σε μια μεγαλύτερη οργάνωση δεν θα χαθεί, δεν θα εξαφανιστεί για να το πω έτσι, απορροφούμενη από ένα μεγαλύτερο οργανισμό και θα πρέπει να έχουμε ειδικέ ρυθμίσεις για τη διαχείριση ε, και τη διοίκηση στο ιστορικό της Europol έτσι ώστε η ΣΕΠΟΛ και η εκπαίδευση να διαφυλάσσεται ως πολύ ξεχωριστή μονάδα και προτεραιότητα για μας της Europol. Αυτά ενημερωτικά λοιπόν για να σας πληροφορήσω για την περισυλλογή αυτή και τον προβληματισμό μας και μας εμπνέει πολύ και η κοινή προσέγγιση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας καλούν όλους έντονα να σκεφτούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες ε, με τέτοιες συνενώσεις και απορροφήσεις μικρών οργανισμών. Ευχαριστώ. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να ε, συγχαρώ τον κύριο Μπάμφη για το έργο του, όσο και την αφοσίωσή του. Αυτό δεν είναι σχόλιο ε, έτσι, ε, εθιμοτυπικό. Ε, είναι αναγνώριση μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Κύριε μέρα συγγνώμη γιατί ο κύριος Μπάνφη ε, ψάχνει τη διερμηνία του και δεν το βρίσκει. Α, τη βρήκε. Λοιπόν, μπορείτε να τα ξαναπείτε. Ε, τίποτα, καλά λόγια έλεγα για σας κύριε Μπαμφή. Σας επενούσα. Ε, εσάς και τη διαχείρισή σας. Και σας λέω, δεν το λέω αυτό από ευγένεια, ε, για φιλοφρόνηση που γι' αυτό ισχύει, αλλά για να αναφερθώ στην αντικειμενική πραγματικότητα. Λοιπόν, από όλα αυτά που σας είπα, ακούσατε ένα τμήμα μόνο. Πρέπει να κάνουμε κάποιο σχόλιο όμως εδώ. Το Κοινοβούλιο δεν θα χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα με τον κύριο Πρίβε ε, που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ακούμε τα ε, αναγκαία και τα νυφάλια ε, Σουάβιτερ μόντο, φόρτιτερ ρε. είμαστε στο κοινοβούλιο, που σημαίνει ότι τα λέμε έτσι πιο μαλακά ίσως, αλλά επί τη ουσία είμαστε εξίσου στεναροί. Ε, μου φαίνεται εμένα ανισχυτικό για το μέλλον της ΕΠΟΛ, αυτό που εσείς ονομάσατε διαδικασία προβληματισμού και περισυλλογής. Ωραία. Να συνεισφέρω κι εγώ στον προβληματισμό των κοινών και την περισυλλογή και πιστεύω ότι σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή ε, ενός ε, μοιραίου ξυλώματος της ΣΕΠΟΛ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει επιτάπητος μια δυνατότητα, ένα ενδεχόμενο που από χέρι εγώ απορρίπτω και το λέω. Απορρίπτω το ενδεχόμενο η ΣΕΠΟΛ να ενταχθεί στην Europol. Πολύ δε περισσότερο τη στιγμή που όλα αυτά ε, δικαιολογούνται υπό τον όρο της εξοικονόμησης πόρων. Αυτό είναι τραγικό για την ασφάλεια. Είναι δυνατόν να συνδέουμε την ασφάλεια με την εξοικονόμηση. Και πώς θα εντάξουμε τις ΕΠΟΡ στη Europol. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πράγμα που εγώ απορρίπτω επαναλαμβάνω, <coughs> αλλά αν γίνει δεκτή ως ε, δυνατότητα θα πρέπει να δώσουμε στη Europol όχι μόνο τα ε, απαραίτητα μέσα για την online εκπαίδευση, για την πρώτερη και την, ε, ε, την εικονική όσο και φυσική παρουσία ε, των φοιτητών, αλλά θα πρέπει να έχει και προϋπολογισμό. Οπότε πόθεν οι οικονομίες, εάν έχουμε το αξίωμα ότι πρέπει να βρούμε τα χρήματα, θα πρέπει να τα βρούμε από εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα μετά από 7 χρόνια από την απόφαση του Συμβουλίου, από το 2005 έχουμε τώρα 12, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα τρόπο να πούμε, και εγώ το λέω ως βουλευτής, ότι στην εκπαίδευση για θέματα ασφαλείας ε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και όχι μόνο αυτό, με ναι, διαφορά, μάλλον σε αντίθεση με τα όσα έλεγε ο κύριος ε, όχι, όχι μόνο γίνεται, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη γίνεται μια εξαιρετική εκπαίδευση. Εγώ λοιπόν τι λέω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, την ε, αξία, πώς να πω, τη γενναιότητα να ε, δούμε κατάματα ε, την ε, κηδεία, την ταφή της ε, σε πόλ στη Europol με το νέο κανονισμό. Και τι θα γίνει με αυτές τις εικονικές τάξεις, τα μαθήματα δηλαδή, όταν είναι μια αστυνομία δημοκρατική, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά πώς θα γίνει τώρα περιστασιακά για να συντονιστούν μέθοδοι, χρόνοι και πρακτικές μέσα από περιστασιακά ευκαιριακά σεμινάρια στη Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικών Υποθέσεων. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομίες χωρίς να καμουφλάρουμε μία πραγματικότητα που μπορεί να είναι ανισχυτική και που σήμερα μας ανακοινώνεται. Δύο ιδέες λοιπόν πρόεδρε. Ιδέα πρώτη. Είναι χρήσιμη σε πόλ και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά. Αποτελεσματική, από το 10, το λένε και οι αριθμοί άλλωστε, και οι οικονομίες που κάναμε και οι συμμετέχοντες, αλλά βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα βλέπει έτσι τα πράγματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ το ερμηνεύω αυτό, δεν ε, είμαι βέβαιος, αλλά για να κάνει οικονομίες ε, ε, προτιμάει απροκάλυπτα να απεμπολίσει ε, μια ουσιαστική δομή εκπαίδευση. το βάζει στη Europol χωρίς να αυξήσει και τον προπολογισμό. Αυτά είναι τα θέματα της ουσία και εγώ το επικρίνω και επίση τα απορρίπτω. Αν, εναλλακτική λύση, Πρόεδρε. Ε, αυτό που σα είπα. Να αναζωογονηθούν οι, οι εθνικές εκπαιδευτικές. Ε, στην πόλη μου έχουμε μια θαυμάσια σχολή ε, αστυνομικών. Και να πω και κάτι για να τα ακούσουν και ο κύριος Μπάνφη και ο κύριος Πρίμπε. Ε, στις εθνικές σχολές η καλύτερη εκπαίδευση γίνεται όχι μόνο στις βασικές σπουδέ, αλλά και στη διαδικασία ε, εσωτερικών προαγωγών. Και, τι εννοώ λοιπόν, ότι θα πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, να πούμε στο κοινοβούλιο τα πράγματα έξω από τα δόντια και κύριε Πρίμπε, νομίζω ότι δεν είστε σε διαδικασία καθόλου ούτε προβληματισμού, ούτε περισυλλογής. Τα έχετε όλα σκεφτεί και τα έχετε όλα αποφασίσει. Και αυτά είναι περίπλοκα τα πράγματα, πραγματικά. Γιατί, διότι έχουμε το πρόγραμμα της Σοχόλμης και το πρόγραμμα δράσης σας. Και θα πρέπει να ε, έρθουμε αντιμέτωποι με την προσαρμογή ε, των αποφάσεων του Συμβουλίου για κάποιους οργανισμούς στο ε, θέμα του συνθήκης της Λισαβόνας. Και η Europol λέτε είναι. Εγώ μπορώ να συζητήσω, να συμφωνήσω ότι θέλετε να κάνω διάλογο, αλλά δεν νομίζω ότι η Europol θα πρέπει να έχει και την αρμοδιότητα της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Ούτε της φυσικής εκπαίδευσης εκεί να είναι παρόντες και να είναι σχολή και πολύ λιγότερο online. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Γκένς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα μετά από την πολύ δύσκολη απαλλαγή του 2010 και μετά από την κακοδιαχείριση του 2008. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι η υπηρεσία ανέπτυξε ένα πάρα πολύ σωστό σύστημα διαχείρισης και επίσης χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα όλα τα καλά λόγια από τον κύριο Πρίμπε τα συγχαρητήρια του προς την ε, υπηρεσία, προς την ΣΕΠΟΛ και τον ε, Δόκτωρα Μπάνφη. Άκουσα ακριβώς αυτές τις απόψεις πριν, ε, πρόσφατα και ξαφνιάστηκα διαβάζοντας την μελέτη αυτή η οποία μόλις ολοκληρώθηκε αυτό τον Απρίλιο, φέτος τον Απρίλιο Διαβάζοντας ε, λοιπόν ε, την ε, σύνοψη αυτής της έκθεσης για τις διάφορες επιλογές που προτείνει, λέει σαφώς ότι δεν μπορεί να, να φανταστεί ένα, τέτοιο είδου συγχώνευσης ή άλλες, άλλες δράσεις κατάρτισης όπως έχουν γίνει από την ΣΥΠΟΛ τα τελευταία χρόνια. Και επειδή τα επίπεδα αποτελεσματικότητας είναι χαμηλά, επίσης δεν προβλέπει τη δαπάνη άλλων κονδυλίων. Γι' αυτό ε, ξαφνιάστηκα με αυτά που είπατε. Έχετε αναθέσει, υπάρχει μια νέα μελέτη η οποία κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα ή έχετε αλλάξει προσέγγιση αυτούς τους λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης μελέτης διότι αυτά τα συμπεράσματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη του Απριλίου. Επίσης, τα κράτη-μέλη δεν υποστηρίζουν αυτή τη συγχώνευση. Το ήλεγξα αυτό με ορισμένους συναδέλφους και από ό,τι ξέρω, τα κράτη-μέλη δεν είναι ε, τα, τα κράτη-μέλη τα οποία υποστήριξαν βεβαίως την ανάπτυξη της ε, ΣΕΠΟΛ ε, και το Κοινοβούλιο υποστήριξε την Ακαδημία βεβαίως. θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα επιχειρήματα τα οποία ξεπερνούν αυτή την πάρα πολύ ε, μειοπική προσέγγιση και ελπίζω αυτούς τους τελευταίους μήνες να έχουν σημειωθεί καινούργιες εξελίξεις και έχω εμπιστοσύνη στα λόγια σας. Είπατε ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος ε, ε, σκέψης, ε, μια περίοδος προσανατολισμού και πιστεύω ότι πράγματι μπορείτε να αλλάξετε τον προγραμματισμό. Και δεν νομίζω ότι αυτή η συγχώνευση, αυτή η πρόταση θα υποστηριχθεί από τα άλλα κράτη-μέλη, από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει εγώ από τις που έκανα. Κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπάνφη για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του στην ε, ΣΕΠΟΛ και έκανε με τα φοβερές προσπάθειες για να ανασυγκροτήσει αυτή την υπηρεσία, διότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και τα οικονομικά της Ακαδημίας ήταν χάλια, αλλά και η εικόνα, το γόητρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά επίσης και την εκπαίδευση. Ο προηγούμενος διευθυντής ε, είχε διακριθεί ιδιαίτερα στον τομέα αυτό και ε, όσον αφορά επίσης και την διαχείριση του προσωπικού. Επομένως σας συγχαίρω κύριε Μπάνφη διότι είστε αποτελεσματικός σε όλα τα επίπεδα και αυτό σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα διότι αρνηθήκαμε την απαλλαγή το 2010 αν δεν κάνω λάθος και ε, φτάσαμε ε, τώρα εδώ, τέλος του 2012 και τώρα βλέπουμε ότι αυτή η Ακαδημία, αυτή η υπηρεσία ε, έχει αλλάξει, είναι, αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητά της, η καλή διαχείριση του προσωπικού και ο κύριος Μπάμφη σήμερα δεν μας το ανήκει, και ο, μάλλον κύριε Πρίμπε, μήπως μας κοροϊδεύετε η Κομισιόν πήρε την απόφαση να συγχωνεύσει τις, ε, τους φορείς. Δεν ξέρετε πώς να μας το πείτε και προσπαθείτε έτσι στα τυφλά να προχωρήσετε. Ε, εγώ να σας πω ότι διαφωνώ πλήρως με την πρόταση της, με την πρόταση της Κομισιόν για πολλούς λόγους. Τώρα μια και ούτως ή άλλως ε, είναι αποτελεσματική και είναι καλά οργανωμένη η Ακαδημία. Από, από 2.300 φτάσαμε σε 5.000 φέτος. Εάν δούμε το δίκτυο ίντερνετ έχουμε 12.000 συμμετέχοντες. Επομένως, μήπως θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε γιατί υπάρχουν τόσα αιτήματα ε, κατάρτισης από πλευράς των κρατών μελών. Διότι εμεί θέλουμε να έχουμε μια υπηρεσία αποτελεσματική. Υπάρχει μια προσδοκία από παντού. Βλέποντας τον προϋπολογισμό επίσης βλέπουμε ότι και εδώ χρησιμοποιείται ε, αποτελεσματικά ο προϋπολογισμός. Η αύξησή του είναι ελάχιστη. Ξέρουμε ότι μειώσαμε και τον αριθμό των συνεδριάσεων. Οι ομάδες εργασίες, οι συνεδριάσεις των του Διοικητικού Συμβουλίου που ε, γινόντουσαν χωρίς να έχουμε ποτέ ε, την, τα τιμολόγια για τις δαπάνες. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Μπάμφη ο οποίος οργανώνει σωστά την υπηρεσία αυτή και τώρα που έχουν γίνει όλα καλά ε, θέλετε να την διαγράψετε. Να την... Και, εντάξει, ούτως ή άλλως και οι Βρετανοί θα επιλέξουν το, την δυνατότητα του opt-out, άρα όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Στην Χάγη επίσης ξέρουμε τι θα γίνει με την υποδοχή τη. Επομένω, δεν υπάρχει διαφωνία. Επομένω, διαρωτώ με γιατί ξαφνικά, ε, ενώ η Κομισιόν ήθελε στην αρχή να ενισχύσει την ΣΕΠΟΛ πριν από λίγο καιρό, ενώ τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ΣΕΠΟΛ, διότι η ΣΕΠΟΛ έχει γίνει πολύ αποτελεσματική και οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου θέλουν να υποστηρίξουν ε, ε, την, ε, την ΣΕΠΟΛ, η, η, η Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ, ε, αποφασίζει ξαφνικά να εγκαταλείψει την κατάρτιση των αστυνομικών, διότι αυτό συνέβη ούτως ή άλλως. Να μας εξηγήσει η κυρία Μάλστρομ τις απόψεις της. Ευχαριστώ κυρία Μόρβαϊ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά και θα ήθελα να ε, καλωσορίσω και στα Ουγγρικά τον κύριο Μπάνφη, το διευθυντή της ΣΕΠΟΛ. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που ένας Ούγγρος εμπειρογνώμων ηγείται αυτού του Ινστιτούτου και χαίρομαι πολύ ε, που η έδρα είναι Βουδαπέστη αυτού του Ινστιτούτου ε, ε, και μάλιστα στο δρόμο Μπούσεριν που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Στην οδό αυτή. Ε, αλλά εντάξει, αυτό δεν σας ενδιαφέρει μάλλον εσάς. Όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στο διαδίκτυο, χαίρονται ιδιαίτερα. Ε, επειδή βλέπουν έναν Ούγγρο εμπειρογνώμονα στην κορυφή της Ευρωπαϊκής ε, Αστυνομικής Ακαδημίας. Δυστυχώς πολύ λίγα μέλη είναι παρόντα και αυτό στην Ουγγαρία το κρίνεται ως λίγαν απογοητευτικό. Η αστυνομική εργασία, η δουλειά των αστυνομικών δεν είναι αποτελεσματική όσο πρέπει και όλοι πιστεύουν ότι επιτέλους θα πρέπει να αποκτήσουμε μια ισχυρή αστυνομία η οποία θα προστατεύσει τους πολίτες από τα εγκληματικά στοιχεία έχετε μειώσει τον προϋπολογισμό κατά 25%. Φαντάζομαι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες χαίρονται ιδιαίτερα γι' αυτό. Εγώ είμαι ποινικολόγος <coughs> και ήθελα να ρωτήσω ότι πώς διεξάγεται η καθημερινή σας εργασία στην Ακαδημία, η καθημερινή ζωή, ε, πώς τα περνάτε δηλαδή και πώς ε, διαμορφώνεται και την κατάρτιση. Αναφέρατε την εμπορία ανθρώπων, την εμπορία γυναικών, ότι αυτό αποτελεί ένα, μια προτεραιότητα στην κατάρτιση, στα προγράμματα κατάρτισης. Πράγματι είναι ένα πολύ λυπηρό θέμα αυτό και για την Ουγγαρία στο, στο, στην κόκκινη γειτονιά, στη γειτονιά των Πορνίων δηλαδή, στο Άμστερνταμ, εκδίδονται πάρα πολλές ανατολικοευρωπαίες ε, και γυναίκες από την Ουγγαρία, που είναι θύματα της ε, σεξουαλικής εμπειρίας, της εμπορίας ε, γυναικών και παράνομης διακίνησης. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, πώς έχετε διαμορφώσει το πρόγραμμά σας για αυτό το πρόβλημα και πώς μπορείτε μέσω της καθημερινής σας εργασίας να μετατρέψετε τους στόχους σε πραγματικότητα. Ο ρόλος των γυναικών επίσης ε, στις ε, διαπροσωπικές σχέσεις, στην οικογένεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο να απασχολεί και το Κοινοβούλιο. Πώς ε, διαμορφώνεται λοιπόν την κατάρτιση σε αυτό το θέμα. Έχετε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα νέα κράτη-μέλη έχουν ορισμένα, μειονεκτούν σε ορισμένους τομείς, διότι υπάρχουν ορισμένες περιφέρειες, αλλά και σε μικρότερες ε, χώρες, όπως στην ε, Νότια Ευρώπη. Υπάρχουν, ας πούμε, ε, άνθρωποι που απασχολούνται στη γεωργία και καθημερινά μάχονται κατά της ζωοκλοπής και άλλων κακών δυσμενών φαινομένων. Η ζωοκλοπή λοιπόν παρατηρείται συχνά. Επίσης ε, διαρρήξεις, ε, διαρρήξεις, ε, κλοπές. Αυτές είναι πράξεις βίας και εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν επιπτώσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ε, πρέπει να, να έχουμε τη δυνατότητα να ζουν οι άνθρωποι αυτοί με ασφάλεια και να μπορούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Το άλλο θέμα επίσης είναι το δικαίωμα του... το 2006. Συνέρχεστε. Και ακριβώς αυτό το συζητήσαμε, το, το είδαμε να εκδηλώνεται με ειρηνικές διαδηλώσει στην ε, Ουγγαρία το 2006 όπου ε, όπου διατέθηκαν παράνομα κονδύλια ε, και διαδήλωσαν κατά αυτόν και συνεχεία είχαμε διάφορες, ε, την παρέμβαση, την επέμβαση μάλλον της αστυνομίας αυτές τις ελληνικές διαδηλώσεις ε, κατά δυσμενή τρόπο. Αναφέρατε ότι η Ακαδημία σας είναι και επιστημονικό όργανο, επιστημονικό φόρουμ. Και στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζουμε να μην δούμε στο μέλλον να επαναλαμβάνονται αυτές οι βίες πράξεις από πλευράς αστυνομία. Ε, αυτή η βιαιότητα δηλαδή η αστυνομία να μην υπάρχει και να μην ξαναδούμε τέτοιες περιπτώσεις ε, στο μέλλον, όπως είδαμε στο παρελθόν. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς διεξάγεται η καθημερινότητά σας στην Ακαδημία σας, ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ε, ε, ε, τότε δίνω το λόγο στην εισηγήτα, η κυρία Μάκιντάιρ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον δόκτωρα Μπάμφη και τον κύριο Πρίμπε που ήρθαν σήμερα το απόγευμα και μας μίλησαν. Με ενδιαφέρον τους ακούσαμε. Ως εκλεγμένο μέλος προτιμώ να συγκεντρωθούμε στους στόχους και ιδιαίτερα στα επιτεύγματα της Ακαδημίας και όχι στον τρόπο που λειτουργεί, που έχει οργανωθεί. Εκεί θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μου. Διαβάζοντας ε, τώρα το σύντομο σημείο, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία δεν είναι ε, ένα, είναι ένας, ε, είναι ένα δίκτυο. Κοιτώ, λοιπόν, στο παρελθόν, α, κοιτάζοντας την Βρετανική νομοθεσία, θα έλεγα ότι εάν ο ορισμός της Ακαδημίας ήταν ένα εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα θα, είχε υποστεί τις διατάξεις του νόμου, τις επιπτώσεις του νόμου περί ψευδών δηλώσεων. Λοιπόν, δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένα δίκτυο. Ε, το, εάν, εάν η Ακαδημία διοργάνωνε ε, προγράμματα για την αστυνόμευση, όχι τόσο για την αστυνομική συνεργασία, Θέλω δηλαδή η αστυνόμευση να είναι το κέντρο βάρους και όχι η δημιουργία περαιτέρω γραφειοκρατικών ε, διαδικασιών, δικτύων κλπ. Ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε εγκληματικές δραστηριότητε. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Ιδίως στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη. Ακριβώς ε, χτες μιλούσαμε για την εμπορία παιδιών ε, και τη τεράστια δυσκολία που υπάρχει υπάρχει, να καθορίσουμε ακριβώς τις συγκεκριμένες διαφορές και να οριοθετήσουμε τις διαφορές μεταξύ ενός ε, ανθρώπου που ζητάει άσυλο και μιας περίπτωσης εμπορίας παιδιών. Ε, αυτά ακριβώς, αυτές τις ενέργειες πρέπει να, να αποτελούν το στόχο μας. Όταν εξετάζουμε θέματα ε, ε, οργανωμένου εγκλήματος, καταπολέμησης εγκλήματος ε, και ξέπλυμα χρημάτων είναι δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Πώς μπορούμε να πώς μπορείτε να στοχεύσετε τις δραστηριότητε σας στα σημαντικά ακριβώς αυτά προβλήματα, στην καταπολέμηση αυτών των σοβαρών ε, εγκλημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος και όχι να διασπάσετε τις ενέργειες σας και να επικεντρωθείτε μόνο ε, στα προγράμματα κατάρτισης και συνεργασίας. Εγώ πιστεύω ότι η καταπολέμηση είναι πολύ καλύτερη από τυχόν απόδοση πτυχίων. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε κυρία Χιμένης ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέμπερ και εσάς κύριε Πάνφη για την παρουσία σας και τις παρουσιάσεις σας εδώ. Θέλω να σας εξηγήσω ότι ως εισηγήτρια της έκθεσης για τα δικαιώματα και τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων αξιόπινων πράξεων που ψηφίστηκε στη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, θέλω να σας πω ότι όταν καταρτήσαμε αυτή την έκθεση, η Επίτροπος Ρέντινγκ, που ενδιαφερόταν πολύ και η ίδια, όπως και εγώ, είπαμε ότι στην Ευρώπη έχουμε 75 εκατομμύρια θύματα εγκλημάτων το χρόνο. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Και αφιερώσαμε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της έκθεσης στην πρώτη επαφή που έχει ένα θύμα εγκλήματος όταν πηγαίνουν στην αστυνομία ε, τα θύματα να καταγγείλουν τι τους συνέβη και ποια είναι η πρώτη τους επαφή με τους αστυνομικούς. Και εκεί έχει σημασία η εκπαίδευση και μιλήσαμε με πολλούς αστυνομικούς και καταλάβαμε ότι δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση ούτε την εκπαίδευση πώς να προετοιμαστούν για να έχουν αυτή την πρώτη επαφή με τα θύματα άλλων χωρών, έτσι, όταν μιλάμε για αυτό το πρόβλημα, ε, είναι διασυνοριακό, ανεξάρτητα από τη χώρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία αυτή ε, και η δική σας αστυνομική υπηρεσία, ε, ακαδημία μάλλον, δεν έχει μεγάλο νόημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία να ψηφίζει. 600 τόσες ψήφους υπέρ είχαμε για την ε, συνεργασία της αστυνομίας, για την εκπαίδευση, για το πώς θα ε, συζητούμε τα θύματα, γιατί είναι θύματα κάθε είδους τρομοκρατίας, διακίνηση ανθρώπων, οργανωμένου εγκλήματος, ανήλικοι, ανάπηροι. Ε, και ε, πάει λέγοντας, όταν μιλούμε για θύματα αξιόπινων πράξεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η ομάδα και θα πρέπει η αστυνομία να γνωρίζει ότι υπάρχουν θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και θα πρέπει και η ίδια νομία να καταλάβει και να ε, δει από την αρχή τι είδους μεταχείριση θέλει το κάθε θύμα. Δηλαδή χρειαζόμαστε καλύτερη αστυνομία με καλύτερη εκπαίδευση και ευρωπαϊκή εκπαίδευση σε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διατηρείται αυτό, όχι μόνο το εθνικό που μπορεί να γίνει ήδη, να το έχουμε ήδη στις χώρες μας. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να μην τα παίρνουμε ελαφρά την καρδία αυτά, αλλά να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τον προβληματισμό, αν προβληματίζεστε ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Χιμένες Μπεσερίλ. Βλέπω ότι έχουμε ολοκληρώσει εδώ ε, το κύκλο των μελών της Επιτροπής που ήθελα να μιλήσουν σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα της ημέρας και προχωρούμε εμείς τώρα με τη σειρά μας ε, και δίνουμε το λόγο στους δύο προσκεκλημένους για να απαντήσουν. Κύριε Μπάμφη. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά κύριο λόγο, αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή είναι πολύ προσωπικό. Το 2010, για πρώτη φορά στη ζωή μου, που μπήκα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και είχα μεγάλα όνειρα. Ε, δηλαδή ένα μεγάλο όνειρο που είχα στη ζωή μου έγινε πραγματοποίηση. Πραγματοποιήθηκε τη στιγμή εκείνο. Εκείνη. Και μετά από την πρώτη ακρόαση από την επιτοπή Υπεύθυνη για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού στεναχωρίσκα. ιδιαίτερα διότι δεν πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου. Δεν ήταν αυτά τα οποία ενερευόμουν, αυτά τα, οποία άκουσα τότε στην πρώτη μου επίσκεψη. Μετά από τρία χρόνια που ξανάρχομαι εδώ. Άκουσα σήμερα ορισμένα καλά λόγια. Αλλά δεν ε, είναι δικιό μου, δεν είναι δικά μου επιτεύγματα αλλά είναι επίτευγμα όλων των συναδέλφων, των 200 συναδέλφων στην Αστυνομική Ακαδημία που δραστηριοποιούνται στις 27, στα 27 κράτη-μέλη και διαθέτουν όλες τους τις δυνάμεις για την αστυνομική κατάρτιση. Αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήριά σας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω αύριο είναι να συμμεριστώ μαζί τους τα καλά σας λόγια και τα θετικά σχόλια. Σαφώς δεν είμαστε τέλειοι. Δεν ήθελα να δημιουργήσω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ξαφνικά γίνεται τέλειο σώμα. Κανένας δεν είναι τέλειος. Και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους εξέφρασαν ε, σημαντικές παρατηρήσεις και επικρίσεις τις οποίες σημείωσα. Ε, οι απόψεις σας ε, προσφέρουν την απαραίτητη εγγύηση για τον έλεγχο που εκτελεί το σώμα Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Και εμείς τις σημειώσαμε και θα τις λάβουμε υπόψη για, στη μελλοντική μας πορεία. Τώρα, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν, το Ευρω... η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία από το 2010 έχει επεξεργαστεί ε, ε, προγράμματα αξιολόγησης της κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά σεμελιώνονται ε, ή μάλλον εκπονούνται σε συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα Κατάρτισης το ε, συμπέρασμα, τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης έδειξαν ότι όλα τα μέλη ε, της, ε, και όλοι όσοι επιτελούν την κατάρτιση είναι εμπειρογνώμενες, είναι εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένα άτομα, εξαιρετικά στελέχη. Η απόφαση που είχε ληφθεί όταν δημιουργήθηκε η Ακαδημία είναι ότι ΣΥΠΟΛ θα πρέπει να λειτουργεί επί τη βάση του Εθνικού Προγράμματος Κατάρτισης των Εθνικών Φορέων. Εμείς χρησιμοποιούμε το προσωπικό και τα στελέχη που είναι διαθέσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν θέλετε να διασφαλίσετε την ευρωπαϊκή διάσταση της αστυνομικής συνεργασίας πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε και να ε, εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας την τεράστια πυρογνωμοσύνη των ε, εξειδικευμένων στελεχών. Είμαστε στα χέρια των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ελπίζω η καινούρια λύση και τα καινούρια στοιχεία νέες εξελίξεις θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο έργο μας ως αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής κατάρτισης και αξιολόγησης μπορούμε να επεξεργαστούμε ορισμένα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης τα οποία στοχεύουν στην ε, διακίνηση ε, ε, και εκμετάλλευση ανθρώπων, στην εμπορία ανθρώπων. Έχουμε αναπτύξει ένα καινούριο πρόγραμμα, ένα καινούριο υλικό με το οποίο θα ε, ε, εκπαιδεύσουμε τα ειδικά στελέχη για αυτό το θέμα, σε εμπορίε ανθρώπων. Έχουμε επίσης και ειδικά προγράμματα όπου καλούμε τους εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν ε, τους ε, εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ε, εμπειρογνωμόνων και στελεχών, έτσι ώστε ε, τα άτομα από τη Γαλλία, εμπειρογνώμονες ας πούμε, να μπορούν να πάνε στην, σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, και από εκεί εν συνεχεία να προσφέρουν την εμπειρία τους ε, από την ε, Πολωνία, ας πούμε, στη Γαλλία. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το, το έγκλημα της ανθρώπινης διακίνησης, της ανθρώπινης εμπορίας έχουμε ειδικά προγράμματα, ειδικά μαθήματα. Κάθε τέτοιο μάθημα έχει μια συγκεκριμένη έμφαση, ένα συγκεκριμένο κεντρικό σημείο, ένα στόχο. Ε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, μας λέει ότι ε, η ΣΥΠΟΛ και με την υποστήριξη των προγραμμάτων της Κομισιόν πρέπει να αναπτύξει σεμινάρια, πρέπει να οργανώσει εργαστήρια, σεμινάρια ε, με και, να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς, ε, η Frontex, η Europol, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όχι μόνο κρατικές και δημόσιες αρχές σας είπα ότι έχουμε 200 στελέχη από 27 κράτη-μέλη. Θέλω λοιπόν, προσπαθώ να σας δείξω ότι διαμορφώνουμε τις δραστηριότητες μας έτσι ώστε να ταιριάζουν στους στόχους μας. Δηλαδή κόβουμε και ράβουμε τις δραστηριότητες μας ώστε να ταιριάζουν στο σώμα το οποίο θέλουμε να ε, εκπαιδεύσουμε. Σχετικά τώρα με τις νέες χώρες, Θέλω να πω κάτι για να αποσαφηνίσω τις προηγούμενες παρατηρήσεις μου. Οι αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό με τις περικοπές που έχουν γίνει είναι δραματικές. Αυτά τα, αυτοί οι κατάρτισης είναι, δεν είναι τέλειοι. Όμως λάβατε υπόψη ότι δεδομένου ότι έχουν γίνει τέτοιες τεράστιες περικοπές κονδυλίων δεν μπορούν να, να βρουν εκπαιδευόμενους, να προσλάβουν δηλαδή ούτε στελέχη και ούτε έχουν εκπαιδευόμενους. Γι' αυτό λόγω των περικοπών αυτών έπρεπε να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας και να κάνουμε μια ανακατανομή των κονδυλίων για να εξασφαλίσουμε ότι τα πιο δύναμα κράτη-μέλη μπορούν να στείλουν αυτά τα στελέχη τους στην εκπαίδευσή μας, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Όσον αφορά τώρα την ε, βία στο σπίτι, έχουμε ένα ηλεκτρονικό, ε, έναν ηλεκτρονικό κύκλο εκπαίδευσης, έχουμε μια εκπαιδευτική ύλη την οποία ε, διαθέτουμε στα, στις 27 χώρες ε, για να ενσωματώσουν την ύλη αυτή στα εθνικά τους προγράμματα. Η, βία, η, η οικιακή βία, η βία στο σπίτι, στην οικογένεια είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως μας απασχολεί και έχουμε ειδικά προγράμματα και η ανδροικογενειακή βία και επίσης υπάρχουν ορισμένες φωνές, ορισμένοι που αμφισβητούν αν η ενδοοικογένειακή βία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κατάρτιση της Ακαδημίας μας, δεδομένου ότι δεν έχει ας πούμε διασυνοριακό, διασυνοριακή επίπτωση. Όμως εμείς επειδή θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το περιλαμβάνουμε. Και επίσης ε, ήθελα να επαναλάβω ότι το δίκτυο δεν, ε, που έχουμε δεν είναι απόφαση της υπηρεσίας. Το, το δίκτυο των εθνικών ε, φορέων κατάρτισης είναι απόφαση των ιδρυτικών πατέρων, των ιδρυτικών μελών της ΣΥΠΟΛ. Η εναρμόνιση του εθνικού συστήματος κατάρτισης υπό την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να επωφεληθεί και να συγκεράσει όλη την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση των 27 κρατών μελών. Αυτή ακριβώς ήταν και η απόφαση η οποία ενέπνευσε τη δημιουργία μας. Υπάρχουν διάφοροι που ε, αμφισβητούν ή ρωτούν, εν πάση περιπτώσει, αν αυτό το δίκτυο είναι ακόμα αξιόλογο, εάν αξίζει να συνεχίσει την ύπαρξή του. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι επαναστατικές αλλαγές δεν πρόκειται περί μεταρρυθμίσεως, αλλά περί επαναστατικών αλλαγών που έχουμε κάνει, που έχουμε καθιερώσει μετά το 2010, θα αποδείξουν την αξία μας. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας, αν παρέλειψα κάτι Ζητώ συγγνώμη και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Μπάνφη, για την απόψη σας που με τόση ειλικρίνεια μοιραστήκατε μαζί μας. Ο κύριος Πρίπε για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να επαναλάβω με τρόπο πολύ σαφή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει λάβει απόφαση Εν πάση περιπτώσει θα γίνει πρόταση και θα αποφασίσει ο νομοθέτης. Δεν είναι λυμένη η απόφαση αυτή. Ε, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο επιτρόπων. Είναι γεγονό αυτό, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε και επιτρέψτε μου να το εξηγήσω και πάλι γιατί μάλλον δεν κατάφερα να το κάνω με το σωστό τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι έχει ληφθεί απόφαση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το πώς θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη διαχείριση των τόσων πολλών οργανισμών που έχουμε τώρα, που είναι πάνω από 30. Και ένα από τα σημεία σε αυτό το μακροσκελέστατο έγγραφο για την κοινή προσέγγιση που και εσείς συναποφασίσατε είναι να προβληματιστούμε για την ανάγκη να μειωθεί ένας αριθμός ε, οργανισμών. Μάλλον μια σειρά ε, ε, οργανισμών και όπως είναι πολύ μικροί αυτοί οι οργανισμοί να εξεταστούν πρώτοι. Γιατί δεν αφορά μόνο τις ε, υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όταν είναι μικρή η ε, ε, οργάνωση και ο οργανισμός και είναι συγκριτικά και ποσοστία μεγαλύτερο το διοικητικό άχθος και το γραφειοκριτικό. και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και μας καλεί άλλωστε η κοινή προσέγγιση να το σκεφτούμε με τρόπο σοβαρό και με ανοιχτό πνεύμα. Τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο και δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι καλούμεθα να προβληματιστούμε ακριβώς όταν έχουμε μια περίπτωση όπου η νομική βάση ενός οργανισμού ε, πρόκειται να ανανεωθεί και ε, στην χάνει η ΣΕΠΟΛ να είναι η πρώτη τέτοια περίπτωση μετά την αναθεώρηση της νομικής βάσης, όπου ανανεώνεται η ε, νομοθεσία. Δηλαδή πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να το σκεφτούμε με τρόπο σοβαρό πράγμα, το οποίο και πράττουμε και είναι φυσιολογικό σε τέτοιες συζητήσεις. Εκείνοι που ασχολούνται περισσότερο με ένα συγκεκριμένο οργανισμό θέλουν να διατηρηθούν οι δομές έχουν. Ενώ κάποιοι άλλοι που βλέπουν μάλλον την ολόκληρη εικόνα, τη θεσμική, τα οριζόντια θέματα, τα εγκάρσια των ευρωπαϊκών οργανισμών για το πώς οργανώνονται και πώς διοικούνται, μάλλον ε, θα συνηγορήσουν υπέρ της ε, συγχώνευσης των μικροτέρων οργανισμών. Αυτό τον καιρό αυτό κάνουμε. Είναι προβληματισμός, είναι ε, περισυλλογή, το σκεφτόμαστε και έτσι θα προχωρήσουμε. Θα καθυστερήσει ε, αυτή η προσπάθεια. Έχουμε αναβάλει την αρχική πρόταση. Ε, δηλαδή δεν θα γίνει φέτος, αλλά λίγο αργότερα. Για να αποφύγουμε τις παρανοήσεις. Όταν μίλησα για οικονομίες, δεν εννοούσα ότι ε, θα περικόψουμε τον προϋπολογισμό της ΕΠΟΛ. Δεν το πρότεινε κανείς αυτό. Απλώς θα συνενωθούν ε, μια μικρότερη δομή με μια μεγαλύτερη και έτσι γίνεται οικονομία στις οριζόντιες ε, δομές. Έχουν γίνει πολύ εντυπωσιακέ ε, ήδη ε, οικονομίες, έκανε ο κύριος Μάνφη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Κάτι άλλο που σας είπα που και πάλι είναι θέμα περισυλλογής. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικά μοντέλα. η εκπαίδευση σε σχέση με άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες, ας πούμε, ε, σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ή να αναγνωρίσουμε ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Frontex, που είναι η υπηρεσία συνόρων, ε, ένα από τα καθήκοντά τους είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν θα γίνει και καμιά φοβερή πολιτιστική επανάσταση εάν η εκπαίδευση της αστυνομίας ενταχθεί στη Europol. Υπάρχει και προηγούμενο, το έχουμε ξανακάνει. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα επιχειρήματα που ζητούν να παραμείνουν χωριστά αυτά. Για όπως σας είπα και προηγουμένως, ό,τι και να γίνει θα κάνουμε την πρότασή μας και οπωσδήποτε θα βασιστούμε ε, και θα έχουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες ότι δεν θα χαθεί ε, ε, η προσπάθεια εκπαίδευσης ε, ε, σε άλλους χώρους όπως είναι το Κέντρο για την Εκπαίδευση για το Κυβερνοέγκλημα. Πρόσφατα έχει ανανεωθεί η νομική βάση για τη Frontex, υπάρχει προηγούμενο και εξ όσων γνωρίζω η Europol έχει αναλάβει ήδη κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το κυβερνοέγκλημα, ας πούμε, πρόκειται να το επεκτείνουν. Αυτά ήθελα εγώ να προσθέσω μόνο για να εξηγήσω ίσω καλύτερα ακριβώς τι σκεφτόμαστε και τι μας προβληματίζει και τι προτιθέμεθα να πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ τον εκτελεστικό διευθυντή της ε, του κύριου Μπάμφη. Ελπίζω ο ευρωενθουσιασμός σας να μην έχει πληγωθεί ε, από τις πολλαπλές ακροάσεις στην Επιτροπή Ελευθεριών. Εμείς ελπίζουμε ε, να έχουμε μεγαλύτερη και αγαστή συνεργασία στο μέλλον. Λοιπόν, η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 27 Νοεμβρίου. 26 λέει εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ.